Dear colleagues, please take your seat. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Yeah, ich möchte Sie heute ganz... Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε την παραδοσιακή μας ε, συνάντηση με τα Εθνικά Κοινοβούλια και ο τίτλος της συνεδρίασής μας είναι «Ίση και αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης». Γιατί δεν λαμβάνει χώρα. Αυτό είναι το σημερινό μας θέμα. Και έχουμε 30 περίπου συναδέλφους από τα Αφρικά κοινοβούλια, από 21 κοινοβούλια και 17 κράτη-μέλη, αλλά έχουμε επιπλέον 9 προέδρους επιτροπών περιβάλλοντος από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων. Η διάθεση του προγράμματος είναι ως εξής. Θα μιλήσουμε καταρχήν για τα απόβλητα αλλά και τα θέματα των υδατήρων πόρων και θα αναφερθούμε και στα θέματα της ομοθεσίας Έχουμε υψηλού επίπεδου εισηγητές. Έχουμε τον κύριο Μακάρνι, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Γαελική στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και έχουμε επίσης τον Επίτροπό μας, τον κύριο Ποτόσνικ, ένα τακτικό καλεσμένο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο να έχουμε την παρουσία σας κύριε Επίτροπε και έχουμε επίσης και την Jackie McGlade η οποία είναι εκτελεστική διευθύντρια του, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος η οποία θα παρέμβει στο δεύτερο μισό της συνεδρίασής μας. έχουμε στην ημερησία διάταξή μας, όπως και εθνικά κοινοβούλια, πολλά νομοθετικά θέματα, τα θέματα εφαρμογής επίσης και υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα του περιβάλλοντος. Εμείς πολλές φορές έχουμε ενώπιόν μας τον κύριο Επίτροπο, αλλά και άλλους και προσκαλεσμένους και κάνουμε συζητήσεις για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί που να είναι αποτελεσματικοί. Αυτό είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνουμε όλο και περισσότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο περιβάλλοντος, ποιότητα αέρος, ποιότητα υδάτων. Όλα αυτά δεν έχουν εθνικά σύνορα. Οι βλάβες προς το περιβάλλον δεν γνωρίζουν σύνορα. Γι' αυτό η πολιτική περιβάλλοντος είναι μια από τις παλιότερες πολιτικές στις οποίες δραστηριοποιείται νομοθετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι πολύ σημαντικό για τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών να μπορέσουμε να κάνουμε σαφές ότι μια πραγματική και λειτουργική πολιτική περιβάλλοντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πραγματική προσθέμενη αξία. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει μας ως Επιτροπή Περιβάλλοντος. Μας ενδιαφέρει επίσης και το θέμα της δημόσιας υγείας Το θέμα μας είναι λοιπόν πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εφαρμογή των ε, νομοθεσιών και των ρυθμίσεων για το περιβάλλον. Είπα ότι θα ξεκινήσουμε με τα θέματα των αποβλήτων και του, των υδατίνων πόρων, αλλά έχουμε και το δεύτερο τμήμα της ημέρα διάταξης, όπου θα σταθούμε στο δίκτυο Natura 2000. Δεν έχουμε επιτύχει όλα αυτά τα οποία θέλαμε να επιτύχουμε στο Natura 2000 Ό,τι έχουμε επιτύχει βέβαια πρέπει να υποστηριχθεί και να εξασφαλιστεί. Και εδώ ο κύριος Λίζε, ο κύριος Κάουχ μπορούν να με ακούσουν. Τα θέματα αυτά λοιπόν θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Η περιβαλλοντική νομοθεσία λοιπόν με την σε συνδυασμό με την εφαρμογή της. Αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μακ Κάρτη, όπως προβλέπετε. Ε, έχουμε συμφωνήσει οι συγητές να μιλήσουν το maximum 10 λεπτά και οι ερωτώντες από τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουν 3 λεπτά χρόνο και θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία αντισφαίρησης κατά κάποιο τρόπο, ερωτήσεις, απαντήσεις. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αναφέρετε όταν λαμβάνετε το λόγο το όνομά σας και το κοινοβούλιο από το οποίο προέρχεστε. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τους συναδέλφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμένα τον ίδιο. Αρκετά είπα λοιπόν και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μακάρντεν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει στα αγγλικά ο ομιλητής και συνεχίζει στα αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σα να έρθω εδώ και να πάρω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Ευρωβουλευτές, συνάδελφοι, κύριε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την εισήγησή μου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Κρότε κυρίω για την πρόσκλησή του και για την εισαγωγή που έκανε. Η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να πετύχει τους στόχους της και τις φιλοδοξίες της, έτσι όπως αυτές καθορίζονται από τις συνθήκες και το κοινοτικό κεκτημένο, εξαρτάται απολύτως από την αποτελεσματική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη. Η καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που έχει να κάνει με περίπου 500 εκατομμύρια πολίτες μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον οι κανόνες για την εναρμόνιση εφαρμόζονται παντού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ δεν υπάρχουν σύνορα στην καταστροφή του περιβάλλοντο. Η ποιότητα του αέρα, η προστασία και η διαχείριση των υδάτων, η διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία του εδάφου, η προστασία τη βιοποικιλότητας, η χορύπανση είναι πράγματα τα οποία μπορούν να προστατευθούν μόνο με ενιαίου κανόνε, ενιαίε προδιαγραφέ που θα εφαρμόζονται σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο η σωστή εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να προσφέρουμε καλή ποιότητα ζωής στις επόμενες γενιές. Βέβαια δεν υπάρχει κανένα λόγο γιατί μια χώρα μέλη να μην εφαρμόζει την νομοθεσία που έχουμε έτσι κι αλλιώ υπογράψει όλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το 7 ε, πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που ονομάζεται ζώντας καλά μέσα στον πλανήτη μας, η πλήρης εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανόνων και κεκτημένου ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια επένδυση για την ανθρώπινη υγεία αλλά και για την οικονομία μας. Είμαστε στα μέσα περίπου της Ιλλανδικής Προεδρίας και μέχρι τώρα έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδο σε θέματα όπως, έχει, όπως είναι η μεταρρύθμιση της κοινή ιωρικής πολιτικής, η Τραπεζική Ένωση, η ανακεφαλαίωση των τραπεζών, η, το πακέτο των δύο νομοθετικών πράξεων, η εγγύηση για τους νέους, η εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τέλος η ενιαία το ενίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Από περιβαλλοντική πλευρά, η Ιρλανδία δουλεύει σκληρά για να προωθήσει την πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ευρώπη μέσω του 7ου προγράμματο πλαισίου. Έχουν υπάρξει πολλέ εξελίξει τα τελευταία χρόνια επίση για να βελτιώσουμε την επιθεώρηση, την εφαρμογή και την ε, θέση σε ισχύ της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η συμμετοχή βέβαια των πολιτών στη διαδικασία αυτή αναφέρεται στη σύμβαση του Άρχου και έχει τεράστια σημασία, γιατί πρέπει να συνειδητοποιεί το κοινό ποια είναι η περιβαλλοντική νομοθεσία και να βοηθάει για την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να συμμορφώνονται όλες οι χώρες με την κοινωτική νομοθεσία. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει βελτιώσει την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων στην ε, όλη διαδικασία, βελτιώνοντας την παρουσία των Εθνικών Κοινοβουλίων στην λήψη αποφάσεων. Η Μικτή Επιτροπή του Κοινοβουλίου μας για το περιβάλλον πρόσφατα υπέβαλε ένα έγγραφο στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου είναι το κόμμα 2012-628 όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον διαφόρων σχεδίων εθνικού και ιδιωτικού χαρακτήρα. Και το κάναμε αυτό γιατί η Μεκτή μας Επιτροπή εκφράζει ανησυχίε όσον αφορά το κόστος, το διοικητικό των διαφόρων προτάσεων, κόστος το οποίο επομίζονται τελικά οι σχεδιαστές. Και σαν αποτέλεσμα των συζητήσεων η Επιτροπή μας κατέληξε σε κάποιες συγκεκριμένες ε, προτάσεις εξετάζοντας αδελφώς το ζήτημα και ζήτησε μεγαλύτερη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Αυτή η νομοθεσία έτσι εξετάστηκε ενδελεχώς από τους ε, πολιτικούς σε εθνικό επίπεδο και μπορεί έτσι να επηρεάσει το όλο αποτέλεσμα. Επίσης επιτρέπει την ανάπτυξη παρετέρω προγραμμάτων αλλά υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν μέρο μια ευρύτερη συζήτηση, στην εποχή μάλιστα που εφαρμόζονται μέτρα λιτότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το κόστος της μη εφαρμογή των ευρωπαϊκών ε, περιβαλλοντικών ε, ρυθμίσεων έχει ακόμα μεγαλύτερο κόστο. Διότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι πιο σημαντική από την προστασία του περιβάλλοντος. Η ισορροπία είναι πολύ λεπτή και σίγουρα αντικατοπτρίζουν και την γενικότερη ανησυχία που εκφράζεται στις συζητήσεις που γίνονται για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Στην ε, Ιρλανδία, το τμήμα για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδίκηση, διάφορες τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία συνέρχονται και έχουν παρουσιάσει παραδείγματα από την Ιρλανδία όπου δεν έχουν συμμορφωθεί αρμόδιοι με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό έχει να κάνει με την αποτυχία της Ιρλανδίας να ενσωματώσει ευρωπαϊκή νομοθεσία στην εθνική της νομοθεσία. Αλλά οι δύο αυτές περιπτώσεις που αναφέρω ευτυχώς έχουν λυθεί μέχρι τώρα και τώρα υπάρχει πλήρη συμμόρφωση στην κοινωτική νομοθεσία. Στην Ιρλανδία έχει αναπτυχθεί και μια κοινοτόμα διαδικασία για την προστασία και την πρόθεση των ρυθμίσεων υπέρ του περιβάλλοντος. Έχουμε φτιάξει μια ομάδα που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας όπου εκπροσωπούνται ε, άτομα από το Ιρλανδικό Τμήμα για το Περιβάλλον, από μη κυβερνητικέ οργανώσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ιρλανδία όσον αφορά την εφαρμογή και την πρόθεση της περιβαλλοντικής κοινωτικής νομοθεσίας. Η ομάδα αυτή έχει σαν ε, κύρια καθήκοντά της να φροντίζει για την επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων όταν τίθεται θέμα ενσωμάτωσης εφαρμογής και θέση σε ισχύ της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Να εφαρμόζει μηχανισμούς διαβούλευσης και επικοινωνίας προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται για κάθε αλλαγή που έχει να κάνει με τη δημιουργία, την τροποποίηση, την ενσωμάτωση, την εφαρμογή, τη θέση σε ισχύ περιβαλλοντικής νομοθεσίας και να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτήν. Για να Επίσης, στόχος της είναι η συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης, συνειδητοποίησης και εντοπισμού νέων ευκαιριών για προγράμματα υπέρ του περιβάλλοντος. Επίσης, διευκολύνει το feedback από μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με το περιβάλλον και το Ιρλανδικό τμήμα για το περιβάλλον, την Ιρλανδική υπηρεσία για το περιβάλλον, προκειμένου να μπορούν να συζητήσουν και να προλαμβάνουν καταστροφή του περιβάλλοντο σε όσο γίνεται νωρίτερο στάδιο. Υπάρχει βέβαια ανάγκη φυσικά να ελέγχουμε την αποτελεσματική εφαρμογή τη περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε μερικέ περιοχέ όμω, δυστυχώ αυτό το θέμα δεν βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα. Οι κυρώσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σίγουρα θα βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα όμω πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, να εκπαιδεύουμε, να διαπαιδαγωγούμε τον κόσμο μα, του πολίτε μα, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον. Αυτή η διαπαιδαγώγηση είναι το κλειδί. Και πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στην συνάντηση των ε, Προέδρων των Επιτροπών για το Περιβάλλον των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα λάβει η χώρα 10 και 11 Μαΐου και αποτελεί μέρος της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ιρλανδικής Προεδρίας. Έχουμε προετοιμάσει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το οποίο θα επικεντρωθεί στην συνοχή της πολιτικής ανάμεσα στην επίτευξη κλιματικών στόχων και την βιώσιμη παραγωγή ενέργειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα υπάρξει και ένα κομμάτι που θα αφιερωθεί στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα. Είναι πολύ υποσχόμενο, θα είναι ενδιαφέρον και ελπίζω να σας δω εκεί πολλούς από εσά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μακάρτη, και τώρα νομίζω μπορούμε να ακούσουμε τον ε, κύριο Ποτόσνικ. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους ε, που εκπροσωπούν τα εθνικά κοινοβούλια να ζητήσουν το λόγο με την κοινή κάρτα. Επίσης για την δεύτερο γύρο των ερωτήσεων έχουμε τις πράσινες κάρτες. Αν θέλετε σηκώστε το χέρι σας με την ε, αντίστοιχη κάρτα για να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τους ομιλητές και να οργανώσουμε την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Στις 5.30 ε, έχουμε προβλέψει ένα μικρό κοκτέιλ έξω από την αίθουσα και βεβαίως ε, είστε όλοι προσκεκλημένοι. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο για το θέμα, το πρώτο θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίας, κύριε Μακάρτη αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους. Είμαι πολύ ευτυχής, διότι μπορώ σήμερα να μιλήσω για ένα θέμα που πραγματικά με αφορά και το οποίο έχει τεθεί σαν προτεραιότητα όσον αφορά την αποστολή μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκύπτει το θέμα της νομοθεσίας. Και βεβαίως εδώ το θέμα που μας αφορά είναι οι επιλογές που έχουν γίνει όσον αφορά την περιβαλλοντολογική νομοθεσία και να δείξουμε το κατά πόσο έχει γίνει πρόοδο στους τομείς αυτούς. Για να μετρήσουμε την πρόοδο πρέπει κανείς να κάνει μια μικρή ιστορική αναδρομή στην αρχή στους πρώτους μας φιλόδοξους στόχους όταν πήραμε τις πρώτες αποφάσεις για το ε, νερό και για τα απόβλημα την δεκαετία του 70, του 80 για την προστασία της δημόσιας υγείας βασιστήκαμε στα πρότυπα όσον αφορά το πόσιμο είδωρ και όσον αφορά τα υδατά κολύμβησης. Ήταν οι πρώτες οδηγίες και βεβαίως ασχοληθήκαμε και με το θέμα των λιμάτων και την επεξεργασία των αποβλήτων. Θα ήθελα την ίδια ώρα να σας πω ότι ήδη από το 2015 έχουμε θέσει τους στόχους και την οδηγία πλαίσιο η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί. Για τα λύματα και τα απόβλητα οι στόχοι μας ήταν εξίσου φιλόδοξοι. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την υιοθέτηση της πρώτης αυτής της νομοθεσίας πλαίσιος και βεβαίως όλα τα λύματα και απόβλητα θα πρέπει να ελέγχονται και να επεξεργάζονται με ένα ασφαλή και ομοιόμορφο τρόπο. Οι στόχοι μας ήταν πολύ συγκεκριμένοι τρόποι επεξεργασίας των κατηγοριών των λιμάτων και των αποβλήτων με μια διασυνοριακή αντιμετώπιση. Το ερώτημα εδώ είναι αν πραγματικά οι στόχοι μας, οι φιλόδεξοι στόχοι μας έχουν αποφέρει αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα βεβαίως ε, είναι κάτι που μπορούμε να το μετρήσουμε όσον αφορά την ε, ποιότητα των υδάτων, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι έχει επιδεινωθεί. Μπορούμε να δούμε παραδείγματο χάρη την οδηγία του 2011 για τα ύδατα κολύμβησης. 92% των υδάτων βρίσκονται στο ελάχιστο, στο χαμηλότερο όριο όσον αφορά την ποιότητα. Βλέπουμε ότι από το 1990 και το 2009 οι στόχοι μας όσον αφορά τις ακτές παραδείγματος χάρη το 20% βρίσκεται σήμερα στην υψηλότερη ποιοτική κατηγορία. Η οδηγία, η αντίστοιχη για τα λίματα, βρίσκεται σήμερα σε ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά δηλαδή τις κατηγορίες που έχουμε θέσει, 77% ανταποκρίνονται στα υψηλότερα στάντη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι αν κοιτάξει κανείς τους χάρτες για την επεξεργασία των υδάτων και των υδάτων κολύβησης, αντιστοιχούν στους στόχους. Επιτέλους, ήθελα να πω ότι τα τελευταία στατιστικά στοιχεία για την επεξεργασία των λιμάτων μας δείχνουν ότι έχει μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων και των λιμάτων και όσον αφορά την ανακύκλωση, από το 27% το 2001 έχουμε φτάσει το 40% το 2011. Βεβαίως όμως αυτό δεν αρκεί. Η δημόσια υγεία, η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στο κέντρο αυτών των προσπαθειών μας και βεβαίως έχουμε διαπιστώσει σήμερα ότι όλες αυτές οι νομοθετικές προσπάθειες θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πιο φουλάδεξους στόχους. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει τους αρχικούς μας στόχους, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Η υλοποίηση βεβαίως μπορεί να μας οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την εξοικονόμηση του άνθρακα και όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η συμμόρφωση όσον αφορά την νομοθεσία για την επεξεργασία των αποβλήτων μας έχει οδηγήσει σήμερα στην εξοικονόμηση της τάξης των 42 δισεκατομμυρίων και θα μπορούσαμε μέχρι το 2020 να δημιουργήσουμε 400 χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης. Όσον αφορά το πόσιμο είδο, την επεξεργασία των υδάτων, η υπηρεσία των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολεί σήμερα 600.000 άτομα. Με νέες ε, εξελίξεις και χρησιμοποίηση των νέων δυνατοτήτων της αγοράς μπορούμε πραγματικά να είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των δάτων. Παρ' όλα αυτά παραμένουν σημαντικά προβλήματα άλυτα και τα νέα στοιχεία μας δείχνουν ότι περίπου οι μισές λεκάνες υδάτων δεν πρόκειται να έχουν φτάσει τους στόχους που έχουμε θέσει για το 2015, στόχους που έχουν τεθεί εδώ και 15 χρόνια. Και τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία για την υλοποίηση βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα σχέδια για την διαχείριση των υδάτων των ποταμών, των λεκανών και την ίδια ώρα διαπιστώνουμε ότι τα σχέδια αυτά, τα οποία είναι καθοριστικά για να διαφυλάξουμε αυτούς τους πολύ χρήσιμους υδάτινους πόρους και να διαφυλάξουμε την ποιότητα των υδάτων. Παραμένουν επίσης προβλήματα όπως ε, τα αστικά λύματα, των οποίων η επεξεργασία εξαρτάται από τη δημιουργία υποδομών. Βλέπουμε ότι τα επίπεδα συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2004 για την επεξεργασία των λύματων είναι πολύ χαμηλά και από 14% έχουμε φτάσει το 39% οι εκτιμήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής φτάνουν περίπου τα 14 δις επενδύσεις για τα επόμενα χρόνια για να φτάσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Οι μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν σήμερα σημαντικές αδυναμίες και μόνο 11 από τις 27 έχουν ολοκληρώσει τις υποδομές. Βλέπουμε επίσης ότι περίπου 37% των ε, δημοτικών αστικών αποβλήτων επεξεργάζονται και συνεχίζουν να υπάρχουν χωματερές, χωματερές οι οποίες δεν ελέγχονται και οι οποίες αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και για, την, για το περιβάλλον. 27, συγγνώμη, 57 διαδικασίες επί συνεχίζονται σήμερα, βρίσκονται εν εξελίξη για τέτοιες ανεξέλεγκτες χωματερές. Τα κράτη-μέλη βεβαίως βρίσκονται σήμερα στην ε, πρώτη γραμμή όσον αφορά την δράση τους για να υλοποιηθεί η υπάρχουσα νομοθεσία που αφορά τις ε, χωματερές. Ξέρετε ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας και συμμόρφωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες που έχει για την ε, συμμόρφωση και την επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας. Υπάρχουν μεγάλες και μικρές περιπτώσεις παραβιάσεων και για τα λίμματα και για τα απόβλητα και πολλές φορές βλέπουμε συστημικά σημαντικά σφάλματα και αδυναμίες. Υπάρχουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η πίεση αυτή βοήθησε και εδώ στις Βρυξέλλες, ενώ βλέπουμε ότι οι υποδομές όσον αφορά την επεξεργασία των λιμάτων βελτιώνονται, κάτι που βέβαια δεν έχει αποφύγει τις ε, διαδικασίες ε, μπροστά στα δικαστήρια. Βλέπουμε ότι η μεταφορά της κοινοτική ε, νομοθεσίας σε πολλές περιπτώσεις στην εθνική νομοθεσία είναι ελλειπής, καθυστερημένη ή ανεπαρκής. Βλέπουμε επίσης ότι ο εθνικός νομοθέτης πολλές φορές καλείται να συμπληρώσει την υπάρχουσα νομοθεσία. Όσον αφορά την, την οδηγία πλαίσιο για το νερό υπάρχουν εννέα διαδικασίες επί παραβάση και βεβαίως είναι αυτονόητο ότι αν δεν υπάρχει σωστή συμμόρφωση με την οδηγία πλαίσιο θα συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιε διαδικασίε. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά που μπορούν να γίνουν είναι πολλέ φορέ περιορισμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρκετά μέσα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλέ ε, ε, προσφυγέ και διαμαρτυρίε. 500 διαμαρτυρίε οι οποίες σήμερα παρακολουθούνται και ελέγχονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Δεύτερον, βλέπουμε ότι οι διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα πρέπει πολλές φορές να συμπληρωθούν, να δικαιολογηθούν, να στοιχειωθούν και αυτό βεβαίως βλέπουμε ότι σήμερα προσκούει σε σημαντικές δυσκολίες όσον αφορά το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό και η Επιτροπή βεβαίως θα συνεχίσει σαν θεματοφύλακα των συνθήκων να παίζει το ρόλο της. Εμείς όμως θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε τις προσπάθειες τον προηγούμενο μήνα. Παρουσίασα εδώ σε αυτή την Επιτροπή το έντυπο για το νερό, water blueprint. Και επιθυμούμε εδώ να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις διμερείς επαφές τους για την υλοποίηση αυτής της νομοθεσίας και την συμμόρφωση την ίδια ώρα. Σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συνεχιστεί η επικοινωνία προς τους Ευρωπαίους πολίτες έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα. Υπάρχει και ο δικός χάρτης όσον αφορά τα 10 κράτη-μέλη που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις χωματερές. Πρόκειται για ξεχωριστές ε, συστάσεις που έχουν δημοσιευθεί όσον αφορά τη συλλογή των αποβλήτων και την ε, σωστή διοίκηση αυτών των υπηρεσιών. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια βεβαίως είναι πολύ σημαντικά και εδώ προσπαθούμε βάσει συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων να επενδύσουμε βάσει της ε, οδηγίας πλαίσιου. Αυτό βεβαίως βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και μιας ιεραρχίας. Θα συνεχίσουμε επίσης να στηρίζουμε με τα κοινοτικά κονδύλια την ε, επεξεργασία των λιμάτων για την περίοδο 2014-2020. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Βεβαίως, το μήνυμα της ε, επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2012 είναι πολύ συγκεκριμένο. Επιθυμούμε για το 7ο πρόγραμμα για το περιβάλλον, το 7ο πρόγραμμα δράσης, να θέσουμε τους ίδιους φιλοδόξους στόχους. Θέλουμε επίσης να υπάρχουν διαδικασίες έλεγχου έτσι ώστε να μην ε, παραμείνουμε χωρίς δράση στους τομείς τους οποίους συνεχίζουν να υπάρχουν αδυναμίες. Γι' αυτό και έχουμε υποβάλει ένα πακέτο προτάσεων. Και η έμφαση που δίνεται σήμερα είναι για περισσότερη διαφάνεια με στόχο να διευκολύνουμε τους, και να εντοπίσουμε τους ε, ελέγχους, τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Η Επιτροπή συζητάμε διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά την διαρθρωμένη υλοποίηση και την καλύτερη ενημέρωση για τα προβλήματα υποδομών που συνεχίζουν να υπάρχουν όσον αφορά την επεξεργασία των λιμάτων. Θα πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία, λύσεις για την επίλυση των προβλημάτων και εδώ και οι πολίτες αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να παρακολουθήσουν την κοινοτική δράση. Επίσης, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε οι εταιρικέ σχέσεις, οι συμφωνίες υλοποίηση θα προχωρήσουν. Η Επιτροπή και τα κρατημέλη θα πρέπει να βρουν τρόπους να συμφωνήσουν για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Οι έλεγχοι, οι εποπτεία όσον αφορά την υλοποίηση και τη συμμόρφωση είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχιστεί. Εδώ χρειάζεται παρέμβαση από μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεχίζουν να υπάρχουν παράνομες χωματερές, πάνω από 20 επαναλαμβάνω διαδικασίες ε, επί προβλήματα στις υποδομές, κάτι που οδήγησε σε 30 διαδικασίες ε, που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασίες επί παραβάση. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχιστούν οι έλεγχοι και καλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η συνεργασία σε εθνικό, τοπικό και κοινωτικό επίπεδο. Θα πρέπει όλοι οι επαγγελματίες, οι δικαστικοί, να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει σε κοινωτικό και εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει την ίδια ώρα οι επιθεωρητές, οι ελεγκτές να συνδράμουν τα δίκτυα των δικαστών σε εθνικό επίπεδο. Εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, μας έχουν απευθύνει πολλές διαμαρτυρίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε διαδικασίες ενώπιον της δικαιοσύνης. Πρέπει να προχωρήσουμε με το νέο πακέτο. Πρώτον, με την υιοθέτηση του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλειών. Στηριζόμαστε στη δική σας βοήθεια. Τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει συγκεκριμένα να στηρίξουν την έκθεση του Κοινοβουλίου του Μαρτίου του 2013. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση αυτού του πολύ σημαντικού ε, γεγονότος και ευελπιστώ να ακολουθήσει μια συζήτηση μεταξύ μας. Ευχαριστώ Γιάννη Ποτόνσκι, Ποτότσνιχ, για την ε, παρέμβασή σας και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να σας υπενθυμίσω βέβαια ποια είναι και η κατάσταση στην, ε, στα δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει συζήτηση με το Κοινοβούλιο, μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για το πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα με τις δημοσιονομικές πολιτικές, αλλά και αυτό, αυτό επηρεάζει και τα εθνικά προγράμματα και την εφαρμογή τους, προγράμματα όπως το live, το θέμα των αποκεντρωμένων φορέων επίσης και κάτι το οποίο μου είναι ιδιαίτερα προσφυλές είναι η συζήτηση για την πολιτική περιβάλλοντος. Και είναι μια πολιτική η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, παρέχει προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει 100.000 θέσεις, θέσεις απασχόλησης εφόσον με την προϋπόθεση δηλαδή ότι εμείς θελήσουμε να εφαρμόσουμε με συνεκτικό τρόπο όλα αυτά τα στοιχεία της πολιτικής περιβάλλοντος. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι για γραφειοκρατικούς λόγους δεν θα μείνει στο περιθώριο η πολιτική περιβάλλοντος, να μην θεωρείται ότι είναι πηγή κόστους μονάχα ή πηγή προβλημάτων και δεν πρέπει να φύγει από την διαπραγμάτευση γιατί είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό ως προεθέμενη αξία και ως ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μπαίνουμε λοιπόν στη συζήτηση. Η κυρία Ρότινιτσκα είναι η πρώτη η οποία θα λάβει το λόγο και είναι η πρόεδρος του, της Επιτροπής Περιβάλλοντος στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Κυρία Ρότινιτσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να σταθώ στα λόγια του κυρίου Ποτεοτσνικ. Είπε ότι, ότι η μεταφορά του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο, η μεταγραφή αυτή λοιπόν των νομοθεσιών, αντιμετωπίζει ακόμα πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ έρχομαι από την Πολωνία. Η Πολωνία αντιμετωπίζει ζητήματα με την μεταγραφή αυτή των ε, ευρωπαϊκών οδηγιών και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η νομοθεσία για τα ύδατα και τα νητρικά άλατα. Κατά τη δική μου άποψη το πρόβλημα είναι το εξή. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα ύδατα και τα οικοσυστήματα της Ευρώπης θα είναι υγιή, θα πρέπει να υλοποιήσουμε τον πρώτο στόχο της οδηγίας αυτής για την ποιότητα των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος αυτός είναι πολύ πολύπλοκος να τον επιτύχουμε για ένα πολύ απλό λόγο. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις υπέρ του περιβάλλοντος έρχονται σε σύγκρουση με τις επιταγές της κοινή αγροτικής πολιτικής. Και είναι κάπως πιο εύκολα τα πράγματα αυτά όταν η γεωργία γίνεται σε βιομηχανικό επίπεδο με μεγάλε αγροτικέ εκμετάλλευσει. Ενώ στην Πολωνία έχουμε ακριβώ το αντίθετο. Έχουμε μικρά αγροτεμάχια, μικρέ αγροτικές εκμεταλλεύσει. Είναι πολύ δύσκολο να τεθούν σε εφαρμογή όλε αυτέ οι ρήτρε για το περιβάλλον σε ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολλέ, αλλά πολύ μικρέ οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να ακολουθήσουν αυτού του κανόνε. Έχουμε τώρα μια εθνική νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των υδάτων, αλλά δυστυχώς αυτή η νομοθεσία δεν ε, συμμορφώνεται με αυτά που απαιτεί η οδηγία για την ποιότητα των υδάτων. Γι' αυτό υπήρξε και η διαδικασία επιπαραβάση κατά της ε, Πολωνίας για μη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από την Πολωνία. η πρόταση μιας νέα νομοθεσία στην Πολωνία για τα θέματα αυτά προσπαθεί να καλύψει το κενό αυτό, προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι θα βελτιωθούν τα σχέδια διαχείριση των υδατήρων πόρων, δεν αποτελεί παρηγοριά για μας. Το γεγονός ότι και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ιδανικού χαρακτήρα η εφαρμογή της οδηγίας, αλλά θέλουμε να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Την κυρία Αφιρινοπούλου τώρα θα δώσω το λόγο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Εκ μέρου τη Επιτροπή Περιβάλλοντο τη Ελληνική Βουλή, σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την πρόσκληση. Θεωρούμε πολύ σημαντική αυτή τη ε, βοήθεια στην ενίσχυση τη συμμετοχή στην συζήτηση και στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντο και Πολιτική. Η Επιτροπή μα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, το οποίο βεβαίω είναι αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού μα δικαίου. Κάθε χώρα έχει τι ιδιαιτερότητέ τη, θετικέ και αρνητικέ. Η Ελλάδα είναι μία από τι πλουσιότερε χώρε σε βιοπικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και βέβαια ανάμεσα σε ευρωπαϊκέ χώρε. Είμαστε περήφανοι κατά το 27 τουλάχιστον τη 100 τη ελληνική επικράτεια να καλύπτεται από περιοχέ του δικτύου Natura 2000. Αυτό είναι ένα ευτυχέ γεγονό για τη χώρα μα, παρόλα αυτά πολλέ φορέ περιορίζει αντί να ενισχύει την ανάπτυξη. Ένα από τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και οι τοπικέ κοινωνίε δεν αντιλαμβάνονται το χαρακτηρισμό των περιοχών τους ως ε, τμήμα του δικτύου Natura 2000 ως ευκαιρία αλλά ως περιορισμό στη δική τους ανάπτυξη και πάνω σε αυτό θα θέλαμε τη βοήθεια περισσότερο της Επιτροπής, των επιστημονικών συμβούλων των οποίων έχετε και βέβαια ενισχυμένα προγράμματα, το Life Plus αλλά και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει έτσι ώστε να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα αλλά και να οδηγήσουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη στο χώρο της ανάπτυξης μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχει δε στη χώρα μας και ένα μεγάλο ζήτημα σε σχέση με την κωδικοποίηση του δικαιωμάτου περιβάλλοντος. Υπάρχουν πολλαπλές επικαλύψεις ε, νομοθετικές για αρκετά ζητήματα και αρκετή σύγχυση δικαίου, η οποία καθιστά ακόμα και τους νομικούς, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι σε θέματα περιβάλλοντος, να βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσον αφορά στον εντοπισμό ακόμα του εφαρμοστέου δικαίου, αλλά και της εφαρμογής από αυτή την άποψη θα χρειαστούμε να κωδικοποιήσουμε περισσότερο το ελληνικό δίκαιο περιβάλλοντος αλλά και από την πλευρά της ε, Ευρωπαϊκ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, ε, Κομισιόν θα θέλαμε ίσως μια περισσότερη προσπάθεια στη βελτιστοποίηση αλλά και στην απλοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος διότι και τα κράτη-μέλη να κωδικοποιήσουν το υπάρχον δίκαιο περιβάλλοντος όταν θα δεχθούν τις νέες προσθήκες του ευρωπαϊκού δικαίου πάλι θα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα των πολλαπλών στρωμάτων δικαίου τα ίδια θέματα. Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα, αλλά και ενδεχομένω και σε υπόλοιπα, στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, πρόβλημα σε σχέση με το cost-benefit ανάλυση, την ανάλυση του κόστους και του ωφέλους που έχουν ενδεχομένως αρκετοί επιχειρηματίες για την εφαρμογή του δικαίου, του περιβαλλοντικού δικαίου. Θεωρούμε ότι λειτουργεί πολύ καλά και εφαρμόζεται το δίκαιο το περιβαλλοντικό όταν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα επ' αυτού, αλλά όχι όταν οι ποινέ είναι τόσο χαμηλέ ώστε να μην μπορεί, να μην υπάρχει κάποιο λόγο κάποιο πραγματικά να εφαρμόσει το δίκαιο περιβάλλοντος από άποψη οικονομική. Υπάρχει και μια σειρά άλλων θεμάτων τα οποία θα ήθελα να πτύξω, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος. Θα ήθελα όμως εν συντομία να πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε, καλά, σε μια καλή πορεία σε σχέση με την αντιμετώπιση των ανεξέλεγκτων χώρων ταφής των απορριμμάτων. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σε σχέση με αυτό όμως παίρνουμε τις αντίστοιχε ε, τις και η Επιτροπή Περιβάλλοντος παρακολουθεί πολύ στενά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όμως θα χρειαζόμασταν περισσότερη μεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας πάνω σε αυτό, καθώς επίσης και νέα χρήματα στην ε, καινοτομία σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων και άλλων μεγάλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι παρότι πραγματικά η ποιότητα του πόσιμου ύδατος αλλά και των υδάτων κολύμβησης στη χώρα μας είναι σε πολύ καλό επίπεδο, υπάρχει μια, ένα έλλειμμα πολιτικής για την προστασία της βιοπικιλότητας στα ύδατα. Η Ελλάδα έχει οι οποίε είναι ιδιαίτερα σημαντικέ και για την Ελλάδα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Μεσόγειο και θα χρειαζόμαστε περισσότερα και καλύτερα προγράμματα σε, θέμα, σε θέματα προστασία των Ποσειδονιών, καθώ επίσης βεβαίω και την άμεση ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείριση. Ευχαριστώ πολύ. Vielen Ο από το Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου είναι ένα μόνιμο θέμα στην Επιτροπή αυτή και αυτό είναι πολύ, το γνωρίζουν και οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Εγώ ήμουνα εννέα χρόνια ε, πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία της νομοθεσίας αλλά τελικά δεν είναι μια εθελοντική διαδικασία η εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου, είναι μια νομική υποχρέωση και πρέπει όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε το ενωσιακό δίκαιο να εφαρμόστε και να εφαρμόστε και με ενιαίο τρόπο. Σε ό,τι αφορά τα σκύβαλα, τα απόβλητα, νομίζω ότι εδώ έχουμε να αποκομίσουμε μεγάλο κέρδος από τα θέματα αυτά. Γιατί, όπως είπε και ο κύριος ε, Επίτροπος, έχει τονίσει την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τα απόβλητα, τα σκύβαλα, ως πρώτη ύλη. Αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, δεν θα πρέπει να καίμε τα σκουπίδια, να τα αφήνουμε σε χωματερές. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αξιοποιήσουμε τα απόβλητα αυτά και όχι να τα ρίχνουμε σε σκυβαλότοπους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση της Ευρώπης και να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη πρώτων υλών για τους υδάτινου πόρους, Είδα στην περιοχή μου ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουν να, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, συμμετοχή των πολιτών, να τους συνειδητοποιήσουμε τη, για τη σχέση που έχει η ποιότητα των υδατήρων πόρων για την ε, ευμάρεια της ε, περιοχής τους και υπήρξε θετική ανταπόκριση. Υπήρξε μία νομοθεσία για την συλλογή στοιχείων για τα, τους υδάτινους σπόρους από την δεκαετία του 1990 που από ό,τι μου είπαν οι πολίτες οδήγησε σε μια χαοτική κατάσταση. Και εδώ είναι το θέμα του τι στοιχεία μαζεύουμε για την ποιότητα των ιδίων, των υδάτων και τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν αυτά τα στοιχεία και όταν πρόκειται για διαμεθοριακές περιοχές και την ποιότητα των υδάτων σε αυτά τα μέρη υπάρχει πραγματικά μεγάλο πρόβλημα για την εφαρμογή των ε, προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Επομένως πρέπει να θεωρήσουμε ότι η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων θα πρέπει να είναι μια από τις πρώτες προτεραιότητες μας μέχρι το 2020. Θα πρέπει μέχρι το 2020 να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και εδώ θα πρέπει να συμμετάσχει και το ενωσιακό επίπεδο. Έχουμε μιλήσει ήδη για προγράμματα εταιρικού χαρακτήρα. Το ερώτημα είναι αν επαρκούν αυτά τα προγράμματα ή αν χρειαζόμαστε περαιτέρω μέτρα εφαρμογής, παρακολούθησης για μένα δεν είναι επαρκή μονάχα αυτά τα θέματα της εταιρική σχέσης δεν αποτελούν εγγύηση ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια πιο αυστηρή και επακριβή εφαρμογή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ο Χέιτ Μερίτ, αν το προφέρω σωστά, από τη Σουηδία τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, Άμερετ. Θέλω να αναφερθώ στα απόβλητα και πιο συγκεκριμένα στα απόβλητα που καταλήγουν στα υδατά. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και άλλες προκλήσεις και θα ήθελα να τα συζητήσουμε λίγο αυτά και από την Σουηδική οπτική γωνία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι θα γίνει και στο μέλλον. Πρέπει να μειώσουμε γενικότερα τα απόβλητα και εκείνα από τα τρόφιμα. Να βγάλουμε το, τα φωσφορικά από την τροφική αλυσίδα. Έχουμε βέβαια νομοθεσία, έχουμε εθνικούς κανόνες, έχουμε και χρήματα στον προπολογισμό για αυτούς τους σκοπούς, αλλά να ποιε για μένα είναι οι πιο σημαντικέ προκλήσει. Πρώτον, η περιφερειακή συνεργασία. Αν δείτε τι γίνεται στη Βαλτική θάλασσα, που είναι μια πολύ ευαίσθητη θάλασσα, γιατί γύρω από αυτήν βρίσκονται πάρα πολλέ χώρε και μάλιστα ορισμένε από αυτέ ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί έχουμε συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τι κοινέ μα προκλήσει. Η Βαλτική θάλασσα είναι αλήθεια ότι είτε πρόκειται από την Αγία Πετρούπολη, είτε πρόκειται από τη Στοκόλμη, σε αυτήν καταλήγουν τα απόβλητά μα. Είναι σημαντικό λοιπόν να μπορεί να υπάρχει τέτοια περιφερειακή συνεργασία για να υπάρξουν αλλαγέ υπέρ του περιβάλλοντο. Μια άλλη μεγάλη πρόκληση που έχει να κάνει με τα ύδατα είναι η αλία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει μια πάρα πολύ καλή απόφαση όσον αφορά την αλληλευτική πολιτική πια. Είναι ευθύνη όλων μας να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια καλή αλλιευτική πολιτική για να είναι βιώσιμη η αλία και να μπορούμε και μακροπρόθεσμα να έχουμε μια θάλασσα με ύδατα υψηλής ποιότητας και βέβαια αλλιευτικά αποθέματα. Ο Βιτσέντσο έχει το λόγο. Από τη Ρουμανία. Δεν είναι παρόν. Δεν ναι, ναι, είναι παρόν. Κύριε Ήρμη. Σας ευχαριστώ. Είμαι μέλος ε, της ε, Βουλής του Κοινοβουλίου της ε, Ρουμανίας και με τον συνάδελφο Σίζαρ Τζάτα. Συμμετέχουμε εδώ στην ε, συνεδρίαση. Έχουμε ήδη προετοιμάσει έγγραφα τα οποία τα έχουμε υποβάλει στην Επιτροπή και αναφερόμαστε ακριβώς στην υγιεινή διατροφή και θα ήθελα να σας πω ότι ακριβώς επειδή μας ενδιαφέρουν το θέμα των χημικών ουσιών που βρίσκονται στις τροφές σήμερα, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα αυτό. Σας έχω υποβάλει όλα τα στοιχεία, όλα τα έγγραφα και θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να τα κοιτάξετε. Σας ευχαριστώ πολύ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει μια σειρά ε, συναδέλφων. Ο κύριος Γεμπραντή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και από τη δικιά μου την πλευρά καλωσορίζω τους φιλοξενούμενους μας εδώ, τους αδέρφους δηλαδή από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το όλο θέμα της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για μένα δεν έχει να κάνει τόσο με τη νομική πτυχή. Έχει να κάνει με το θέμα της ε, νοτροπίας. Γι' αυτό είναι πολύ καλό που βρισκόμαστε μαζί εδώ, Ευρωπαίοι και Εθνικοί Βουλευτές, να συζητήσουμε αυτό το πρόβλημα που είναι πολιτικό και όχι νομικό. Εδώ μιλάω βέβαια ως Ευρωβουλευτής. Όταν ε, μιλάω με τα κράτη-μέλη, με ποιον μιλάω, με το Συμβούλιο μιλάω. Και πίσω από τις πλάτες βέβαια του Συμβουλίου υπάρχουν 27 χώρες. Το Συμβούλιο όμως εκπροσωπείται από την εκπεριτροπής Προεδρία. Και αυτή δεν πρόκειται να σχολιάσει για τις θέσεις των επιμέρους χωρών μιλών. Το Συμβούλιο δηλαδή έρχεται και μου λέει ποια είναι η θέση του Συμβουλίου συνολικά. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο σε εμά τους Ευρωβουλευτές να εντοπίζουμε τα πολιτικά ζητήματα που τίθενται από την κακή ή ελλειπή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στις χώρες μέλη. Και γι' αυτό πολύ συχνά στρεφόμαστε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο θεματοφύλακας των ε, συνθήκων και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει για την εφαρμογή ή εν πάση περιπτώσει να στείλει ε, αυστηρές επιστολές στις χώρες μέλη προκειμένου αυτά να συμμορφωθούν και να θέσουν σε εφαρμογή την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αλλά αυτή είναι μια πολιτική λύση για πολιτικά ζητήματα. Η πραγματική λύση όμως είναι συνδυασμός πολιτικών δυνάμεων, από πλευρά δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και έτσι η ερώτηση κατά κάποιο τρόπο που έχω να κάνω εγώ δεν απευθύνεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο στους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ρωτάω λοιπόν, εσείς πόσο συχνά ρωτάτε τους ε, υπουργούς για την εφαρμογή της κοινοτική νομοθεσίας. Γιατί εδώ έχουμε ένα ζωτική σημασία πρόβλημα. Το άλλο που διαπιστώνουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών είναι ότι έχουμε υπουργούς ή επιμέρους χώρες μέλη που μας έρχονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητάμε μαζί τους για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στις διάφορες χώρες. Ποια είναι λοιπόν η γνώμη σας το να καλούμε εμείς ε, υπουργού από τις χώρες μέλη βουλευτές να έρχονται εδώ. Συμφωνείτε? Σας παρακαλώ τηρήστε το χρόνο ομιλία σας γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο κατάλογο ομιλητών. Σίζερ Τζότα από τη Ρουμανία. Ήδη τον ανακοίνωσε ο συνάδελφός του. Το όνομά μου είναι Σίζαρ Τσιώτα. Είμαι μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ρουμανικού Κοινοβουλίου. Δεδομένης της εμπειρίας της χώρας μου για θέματα διαχείρισης ε, των ε, υδάτων σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο, η ολοκληρωμένη πολιτική προσέγγιση σε θέματα βιομηχανίας, γεωργίας μας έχει οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη πολιτική από το αρμόδιο Υπουργείο. Έχουμε μια επιτροπή η οποία σχεδιάζει... Αυτά βασίζονται στον εντογραφικό χάρτη που έχει δημιουργηθεί από τη Ρουμανία και αυτό έχει γίνει σε συνεννόηση με τους, ε, με τους ε, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες, προκειμένου να πιστούν αυτές ότι είναι προς το συμφέρον τους να έχουν καλή πολιτική αποβλήτων. Ανακύκλωση και ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την πρωτοβουλία τους για μια αποτελεσματική Ευρώπη όσον αφορά την χρήση πόρων. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική δάτων. Δεν έγινε το ίδιο. Μόνο το 2004 ετοιμάσαμε την κατάλληλη δίκηση που να ασχολείται ειδικά με τα υδάτα και με την προβληματική των υδάτων. Άρα δεν ήταν έτοιμοι έγκαιρα να συνεργαστούν και με τον ιδιωτικό τομέα. Εδώ μένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Κάποιο μίλησε για τη διασυνοριακή συνεργασία και είπε ότι είναι ζωτική σημασία. Ε, πράγματι, και εμεί εκεί μπορούμε να κάνουμε περισσότερο από ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα. Τέλος, εάν θέλουμε να σεβόμαστε τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, ακόμα και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, τότε θα πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ένα άλλο μέτρο. Θέλω να πω ότι το ΕΠ το καθάριστο χώριο προϊόν δεν είναι το καταλληλότερο για να μετρηθεί η ευημερία των ανθρώπων, γιατί η ευημερία των ανθρώπων εξαρτάται και από ένα περιβάλλον ποιότητος. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται μια, αν όχι παγκόσμια, τουλάχιστον ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Επίτροπε, πείτε μας πού βρισκόμαστε από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βόντε. Θα σας ε, δώσω τη δυνατότητα να απαντήσετε στις ε, πολλαπλές ερωτήσεις που σας έγιναν από τους συναδέλφους. Θα προσπαθήσω. Ίσως ξεκινώντας θα κάνω μία παρατήρηση γιατί είναι τόσο σημαντικά αυτά τα θέματα για την Ευρώπη, για σας, για μας. Κάποια από αυτά που συζητούμε. Πράσινη οικονομία, γιατί έχουν τόσο μεγάλη σημασία όλα αυτά και από την άποψη την περιβαλλοντολογική αλλά και οικονομική για να βγούμε από την κρίση. Αν κοιτάξει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνει ότι πρόκειται για σημαντικό εισαγωγέα ενέργειας. Κοιτάξτε παραδείγματο χάρη αυτή τη στιγμή τις εισαγωγές και τις εξαγωγές εξάγουμε κυρίως ε, υπηρεσίες, αγαθά και εισάγουμε οτιδήποτε αφορά την ενέργεια, τους φυσικούς πόρους. Και για τα επόμενα χρόνια βλέπετε ότι η Ευρώπη εξαρτάται και θα συνεχίσει να εξαρτάται από αυτές τις εισαγωγές στους φυσικούς πόρους και την ενέργεια. Η υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενέργεια μας έχει δώσει αυτά τα στοιχεία. Αυτή η εξάρτηση θα αυξηθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη είναι υψηλότερο από αυτό των πολιτειών και από τις Κίνες βεβαίως και εισάγουμε πολύ περισσότερα από αυτά που εξάγουμε. Έξι φορές περισσότερες πρώτες ύλε. Αν προσθέσει κανείς σε αυτό, αυτό που έχει ξεκινήσει από την αρχή του αιώνα, οι τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας αυξάνονται. Οι εκτιμήσεις είναι ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Καταλαβαίνετε ότι η εξέλιξη αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην βιομηχανική μας πολιτική. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Εάν δεν το λάβουμε υπόψη μας θα έχουμε σημαντικές δυσκολίες στο μέλλον και δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι δομές μας σαφώς και θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτά τα δεδομένα. Χρησιμοποιώντας λοιπόν σήμερα τεχνικές όπως την ανακύκλωση, χρησιμοποιώντας μια οικονομία που θα βασίζεται στην ορθή χρήση, οικονομική χρήση, στη μείωση της πατάλης, στην αποτελεσματική χρήση. Πώς θα γίνουμε λιγότερο εξαρτώμενοι σαν Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι ένας από τους πόρους που διαθέτουμε είναι η δυνατότητα να οδηγηθούμε προς ε, καινοτομία, είναι το μυαλό μας αν θέλετε και πρέπει να κατευθυνθούμε προς μια κατεύθυνση η οποία θα μας οδηγήσει σε περισσότερη ανταγωνιστικότητα. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύσουμε το περιβάλλον. Αυτή λοιπόν η οικονομική, αν θέλετε, προσέγγιση θα πρέπει σαφώς να μας οδηγήσει στη διαπίστωση ότι δεν έχουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό και πραγματικά πρεσβεύω αυτήν την ε, κυκλική οικονομία, αυτήν την ορθή χρήση των φυσικών πόρων που διαθέτουμε. Επανέρχομαι τώρα σε αυτά που με ρωτήσατε. Θα ξεκινήσω με τα νητρικά άλατα, το νερό. Είναι η ερώτηση του Πολωνού συναδέλφου, η πρώτη ερώτηση. Αυτό που προσπαθώ να πετύχω είναι να έχουμε συνοχή στις πολιτικές μας. Η γεωργική πολιτική είναι συνδεδεμένη με την προστασία του περιβάλλοντος. Σήμερα πληρώνουμε αγρότες, τους γεωργούς, για να μην μολύνουν το περιβάλλον και όχι απλώς και μόνο για να μην παράγουν. Σήμερα οι δάτινοι πόροι, εάν συνεχίσουν να μολύνονται, θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε τα κονδύλια τα οποία διαθέτουμε. Καταλαβαίνετε γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία πολλαπλή συμμόρφωση όσον αφορά την νομοθεσία ε, του νερού, αλλά όχι μόνο. Όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να τα προετοιμάσουμε ορθά και με καλή συνεργασία μεταξύ μας. Εάν δεν συνεργαστούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μία οδηγία, όπως παραδείγματος χάρη αυτή για τα νητρικά άλατα, η οποία θα απαγορεύσει. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο πρεσβεύω η προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι μια πολιτική που θα ακολουθείται από θετικές προτάσεις. Όλοι θέλουμε να διαθέτει η Ευρώπη ε, καθαρό πόσιμο νερό. Όσον αφορά το Natura, νομίζω ότι θα ασχοληθούμε καλύτερα στη δεύτερη σειρά ερωτήσεων με το θέμα αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε για το περιβάλλον και αν κάποιος αναπτύξει νομοθεσία για τα επόμενα 50 χρόνια βεβαίω χρειάζεται κωδικοποίηση. Υπάρχει πρόβλημα για την κωδικοποίηση σε πολλά κράτη και για όσον αφορά τα οικοσυστήματα. Μιλήσατε επίσης για τα κονδύλια. Είναι πολύ σημαντική η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα χρηματοδότησης ε, σε εθνικό επίπεδο για το νερό παραδείγματος χάρη. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του το κόστος, το οποίο βεβαίως είναι κόστος και περιβαλλοντολογικό, αλλά και ενσωματωμένο κόστος. Πολλοί αναφέρθηκαν στο σημείο αυτό. Είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό να δούμε το θέμα της φορολόγησης των χωματερών, της καύσης των αποβλήτων με σκοπό να μειωθεί το κόστος από τους άλλους τομείς. Πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε κίνητρα τα οποία θα οδηγήσουν την οικονομία προς κάποιους τομείς. Ο γιο έφυγε, σημείωσα όμως αυτά που ε, ήθελε και θα τα ελέγξουμε. Ο συνάδελφος από τη Σουηδία, νομίζω ήταν πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σας. Όντως έχουμε στόχους για τα απόβλητα, οι οποίοι θα ενημερωθούν, θα προετοιμάσουμε μια πρόταση φέτος για τα είδη διατροφής, μια επικοινωνία προετοιμάζεται και επεξεργαστόμαστε βεβαίως και την ε, επαναχρησιμοποίηση των υδάτινων πόρων. Αυτό ήταν, αν θέλετε, ένα από τα δύο κενά της νομοθεσίας για το είδωρ που δεν είχαν καλυφθεί. Μακροοικονομική προσέγγιση των περιφερειών, μιλήσατε για τη Βαλτική. Είναι, αν θέλετε, μια ενδιάμεση δυνατότητα διαχείρισης σε επίπεδο μεταξύ των ε, κρατών, αν θέλετε, διασυνοριακό. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λυθούν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια περιφέρεια, όπως ε, θέματα που αφορούν τη γεωργία στη βαλτική περιοχή. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μεταξύ των κρατών μελών που μοιράζονται αυτήν την ε, περιοχή. Οι βαλτικές χώρες. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό που είπατε και συμφωνώ όσον αφορά την κοινή πολιτική αλίας όλα αυτά που έγιναν εδώ ήταν πάρα πολύ αξιόλογα. Η πρόταση που αφορά τα κράτη-μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, θέσατε πολύ σωστά ερωτήματα. Ακριβώς αυτά πρέπει να συζητήσουμε. Με ποιο τρόπο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε θέματα τα οποία ό,τι και να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούν να βρουν λύση αποτελεσματική. Όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, είναι σημαντικό να καταλάβει κανείς αυτό που σας είπα στην αρχή. Βεβαίως υπάρχει οδηγία, πλαίσιο για τα απόβλητα, που αναφέρεται στην ιεραρχία των αποβλήτων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει λοιπόν να προετοιμάσουν τα εθνικά του σχέδια για να αποφευθεί η ανακύκλωση. Και τέλος βεβαίως κάτω-κάτω η καύση των αποβλήτων και οι χωματερές σαν τελευταία λύση, ίστατη λύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν ε, λύσεις, απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη πολύ σημαντικά οικονομικά εργαλεία που έχουμε, να σας βοηθήσουμε, να σας στηρίξουμε, να υλοποιήσετε τους στόχους. Η ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων, η επιλεκτική και βεβαίως η δημιουργία κινήτρων έτσι ώστε αυτό να γίνει μια ελκυστική οικονομική δραστηριότητα. Αυτά, αν επιλεγούν τα σωστά κινήτρα, μπορεί να δημιουργήσουν μια δυναμική δημιουργία κινήτρων, η δημιουργία ελκυστικών, αν θέλετε, προϋποθέσεων δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι ζωτική συμμαχία και θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Γεωργικά περιβαλλοντολογικά σχέδια. Λιγότερα χρήματα αλλά όχι τόσο πολύ λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί κάποια από αυτά τα θέματα θα καλύπτονται από τον πρώτο πυλώνα. Επομένω θα έχετε περισσότερο περιθώριο λοιπόν στο δεύτερο πυλώνα. Αυτό το οποίο δεν ε, εκτίμησα είναι η θέληση του Συμβουλίου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ των δύο πυλώνων, το οποίο ανοίγει τις πύλες σε προβλήματα. Παρακαλώ, αφήστε να είναι άθικτος ο πυλώνας αυτός, γιατί με τον τρόπο αυτό, ο δεύτερος πυλώνας, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό το οποίο αναφέρατε. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό <clears throat> τα ποσά αυτά στο δεύτερο πυλώνα να χρησιμοποιηθούν με σόφρονα τρόπο. Τώρα ο Κρίς νομίζω έθεσε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι ένα ετήσιο συμβούλιο περιβάλλοντος για την εφαρμογή θα ήταν καλή ιδέα. Δεν ξέρω πώ θα το αντιμετωπίσει το Συμβούλιο σαν πρόταση, κάτι το οποίο όμω το οποίο εμένα θα με ενδιέφερε γιατί συζητάμε την ποιότητα των υδάτων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περνάμε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση για την ποιότητα των υδάτων, για ορισμένε ουσίες που είναι η προτεραιότητά μα, Ναι, Τελείωσε, τελείωσε αυτή η διαδικασία. Ωραία. Ρίτσαρντ, εσύ ξέρει καλύτερα πόσο δύσκολα ήταν αυτά τα θέματα και πόσο δύσκολο είναι να μπορέσει κανεί στην πράξη να πετύχει κάτι το οποίο καταρχήν το συμφωνούμε όλοι μας. Αυτά είναι τα καλύτερα νέα σήμερα το απόγευμα γιατί είχα υπαλλακτικά και εναλλακτικά σχέδια στην τσέπη μου αλλά δεν χρειάζεται να τα εφαρμόσω. Και για το συνάδελφο από τη Γερμανική Bundestag. Εσεί αναφερθήκατε σε πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία ανέφερα και εγώ στην παρέμβασή μου. Ακριβώς αυτά κάνουμε, Απλώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να καλύψουμε όλα αυτά τα ζητήματα. <clears throat> Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει καταρχήν να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη και εργαζόμαστε για αυτή την πρόταση εφαρμογή που θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευθυγράμμιση των απαντήσεων που δίνουν τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό θα πάρει κάποιο από το βάρο στου δικού μα όμους σήμερα και θα υπάρξει και μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών μελών. Χωρί αμοιβαία εμπιστοσύνη έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Χρειάζεται εμπιστοσύνη μεταξύ κυβερνήσεων και εμπιστοσύνη από του πολίτε τη κυβέρνηση. Για την οδηγία για τα εδάφη έχουμε βέβαια διαφορετικές απόψεις. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρώπη. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Γερμανία είναι αντίον αυτή, γιατί η Γερμανία είναι η μόνη χώρα ή μια από τι λίγε χώρε που τα καταφέρνει πολύ καλά με την ποιότητα των εδάφων και επομένω αυτό θα μείωνε την δουλειά που θα πρέπει να κάνετε εσεί, ενώ συγχρόνω θα εξασφαλίζετε ίσε συνθήκε ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη και εξάλλου η βιομηχανία σα είναι πολύ πιο δυνατή στο να αποκαθιστά την ποιότητα των εδαφών. Και πάλι εσεί θα κερδίσετε στον τομέα αυτό αλλά αν αυτό θεωρείτε ότι θα κάνει πιο δύσκολη τη ζωή σας, το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια πηγή αντίστασης. Θα προσπαθήσουμε και στο μέλλον να σας πείσουμε και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Δεν θα μπω τώρα για όλες τις λεπτομέρειες, αλλά αν έχουμε κάτι το οποίο υπάρχει σήμερα γιατί δίνει τις απαντήσεις η αγορά θα μπορούσαμε να ε, μειώσουμε κατά 20 με 50% το νερό το οποίο χρησιμοποιούμε. Δεν πρόκειται τώρα να σταθώ στο, στη λειτουργία των ντους και αυτά τα θέματα, αλλά ξέρω ότι έχετε κάποιες αρνητικές εμπειρίες και αν υπάρχει ένα πρόβλημα είτε είναι πραγματικό είτε είναι κάτι το οποίο είναι μονάχα στην ανθρώπινη αντίληψη, το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Δεν μπορούμε να περάσουμε κάτι που δεν γίνεται αντιληπτό ως λύση. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Κάποιες χώρες βέβαια ε, το κάνουν αυτό ήδη. Ο συνάδελφος από το Φλαμανδικό Κοινοβούλιο η δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς πράγματι πρέπει να τα αναπτύξουμε αυτά και κάνετε πολύ σωστές παρατηρήσεις. για τα συστατικά και την, ε, αυτά που βρίσκονται στην αρχή του κύκλου ζωής της. Και επίσης ένα συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε στην ε, αδυναμία υλοποίησης κάποιων ε, επιταγών λόγω των μεταβατικών περιόδων. Πολλά κράτη-μέλη πολλές φορές αρχίζουν να βλέπουν το πρόβλημα μόνο όταν τελειώνει η μεταβατική περίοδος. Και αφού έχουν αφήσει κατά μέρο όλα αυτά τα προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε ορισμένε περιπτώσει δεν έχουν εκμεταλλευτεί καν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η οποία είναι διαθέσιμη για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά. Εγώ είμαι βέβαια εδώ για να εξασφαλίσω ότι θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, αλλά οι μεταβατικές περίοδοι είναι αυτές που έχουν αποφασιστεί όχι για να μην εφαρμόσουν νομοθεσία τα κράτη-μέλη, αλλά για να μπορούν να προχωρούν σιγά-σιγά προς την συμμόρφωση. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ λοιπόν την συνέχιση της μη συμμόρφωσης. Επίσης, ένα ερώτημα για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ γειτονικών χωρών. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Το ανέφερε ένα συνάδελφος από την Εσθονία και γι' αυτό ασχολούμεθα επίσης. Ο συνάδελφος από την Πορτογαλία είπε μην ασκείτε πίεση, αλλά πείστε τα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο κάνουμε εμείς από την αρχή. Υπάρχει όμως κάτι το οποίο δεν γίνεται ιδιαίτερα κατανοητό. Αν νομίζετε ότι εμείς θα λαμβάνουμε υπόψη όλα αυτά όταν αναπτύσσουμε, όταν αναπτύσσουμε το κεκτημένο, ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών, κάνετε λάθος. Γι' αυτό έχουμε και κάποιες μεταβατικές περιόδους, ώστε η κάθε χώρα να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει και που τους, τις εμποδίζουν να εφαρμόσουν το κεκτημένο. Και αυτό πρέπει να γίνεται στην αρχή, όχι στο τέλος. Όταν έχει εγκριθεί νομοθεσία, εγώ ως Επίτροπος είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το οποίο με υποχρεώ να κάνω οι κανόνες. Για το παγκόσμιο επίπεδο, συμφωνώ ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ενεργοί σε διεθνέ διεθνές επίπεδο και πράγματι συμβαίνει κάτι τέτοιο πιστεύω. Και Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Ε, η συνάδελφος από την Αυστρία το έθεσε το θέμα αυτό. Αν πηγαίνω, όταν πηγαίνω σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, εγώ ε, θέλω να έχω και μια συζήτηση μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Αυτό που λέτε όμως είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο συστηματικό τρόπο να το κάνουμε αυτό και να υπάρχει μεγαλύτερη συναντήληψη στα κοινοβούλια και έτσι ο ρόλος αυτός των κοινοβουλευτικών μπορεί να είναι πιο εποφελής και να είσαστε πιο ε, καλύτερα εξοπλισμένοι για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε δράση. Επομένω, η έκκλησή σας είναι κάτι το οποίο λαμβάνει υπόψη και τέλος για τον συνάδελφό μας από το Λουξεμβούργο το να ξεπεράσουμε το ΑΕΠ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εργαζόμαστε ήδη γι' αυτό. Ξέρουμε ότι αν δεν γίνει σωστά η παροχή πληροφοριών και αναφορών για τους εθνικούς λογαριασμούς και για την διάρθρωση του ΑΕΠ, τότε η λήψη αποφάσεων από μια κυβέρνηση, η απολύπτη αποφάσεων δεν γίνεται σωστά. Εργαζόμαστε λοιπόν για να έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Κάποιες φορές τα πράγματα πηγαίνουν πιο αργά από ό,τι θα θέλαμε. Η ελπίση μου είναι Βλέπω τον ΟΣΑ, βλέπω την Παγκόσμια Τράπεζα, όλους να κινούνται προς την κατεύθυνση δικτών που ξεπερνούν το ΑΕΠ και <clears throat> ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πάνε τα πράγματα πιο αργά από ό,τι ήθελα, αλλά είναι μια νέα κατεύθυνση η οποία είναι αναπόφευκτο να είναι και η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε. Μακρηγόρησα, αλλά ήθελα να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Γιάννος. Νομίζω ότι αξίζει τα χειροκροτήματα όλων. Είσαστε ένας επίτροπος, τον οποίο με μεγάλη χαρά έχουμε πάντα μαζί μας, γιατί απαντάτε όλα αυτά τα ερωτήματα με μεγάλη ακρίβεια και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμούμε ιδιαίτερα στις ε, ανταλλαγές απόψεων και επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγετε, σας ευχαριστώ που είχατε την ευκαιρία και είχατε το χρόνο, δώσατε στον εαυτό σας τον χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό και μαζί μας και με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Δεν μπόρεσα να δώσω δυστυχώς το λόγο σε όλους, αλλά νομίζω ότι στο δεύτερο τμήμα της συζήτησης αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο και κάνω μια διακοπή πέντε λεπτών και στη συνέχεια θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης που έχει να κάνει με την νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος. Αν θέλετε να καθίσετε όλοι μπορούμε να ξεκινήσουμε την ε, συνεδρίαση για να έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε και με την Jacqueline McLeod. Λέγομαι Καρλ Σλούτερ, εκπροσωπώ, αντικαθιστώ μάλλον τον ε, πρόεδρό μας, ο οποίος αποσιάζει πρόσφατα, ε, προσωρινά. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο σημείο που είναι η νομοθεσία για την προστασία τη κρίση και έχω δίνω το λόγο στην κυρία Μακλέτ που είναι εκτελεστική διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ να μιλήσω μαζί σα. Κυρίω τμήμα του έργου του φορέα μα είναι να μπορέσει να δει πώ γίνεται και η εφαρμογή των πολιτικών από τη στιγμή που έχουν αποφασιστεί και αναφέρθηκε το θέμα της, ε, του να κατανομάσουμε και, να επωνυδίσουμε, εμείς θέλουμε και να δοξάζουμε αυτούς οι οποίοι τα κάνουν καλά και όχι μονάχα να επωνυδίσουμε. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι πιο θετικός τρόπος από το να έχουμε ένα βαθμολόγιο και μονάχα, αλλά σίγουρα μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα με το να προβάλλουμε αυτούς οι οποίοι είναι καλοί στην εφαρμογή. Δεν χρειάζεται μονάχα με το ρόπαλο δηλαδή να υποχρεώνουμε τον κόσμο. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω σήμερα το απόγευμα είναι όμως να σκεφτώ μαζί σας για την προστασία της φύσης σε ορισμένες χώρες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο καλύπτεται από νομοθετικά εργαλεία τα οποία έχουν λιγάκι διχαστικό χαρακτήρα, ενώ αλλού είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο συνένεση. Η νομοθεσία για την προστασία τη φύση είναι κάτι το οποίο έχουμε για πολλά χρόνια πάνω από 20 χρόνια. Έχουμε την οδηγία για τα ενδιατήματα, για τα πτηνά, αλλά και την Natura 2000. Αυτή είναι η σπονδυλική στήλη αυτών των θεμάτων που για μας είναι η προστασία της φύσης. Και το... τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει δεν είναι τόσο θετικά. Είδαμε να υπάρχει σε μεγάλο βαθμό μια αντιμετώπιση στεγανοποίησης. Δηλαδή βλέπουμε τις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις χωριστά τη μία από την άλλη. Επομένως το νέο σχέδιο δράσης μέχρι το 2020 όταν το αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς αυτά τα στοιχεία νομοθεσίας συναρμόζονται μεταξύ τους και με τις άλλες κατατομείς πολιτικές. Αυτό που θέλω να αντιμετωπίσω λοιπόν είναι το πώς σε εθνικό επίπεδο <clears throat> θα τροποποιηθούν αυτές οι προκλήσεις έναντι αυτού που είχαμε στο παρελθόν. Είναι προβλήματα επίμονα, είναι προβλήματα τα οποία είναι πολύπλοκα, είναι προβλήματα που δεν επιδέχονται απλές λύσεις και χρειάζονται ίσως συμμετοχή διαφορετικών εμπλεκομένων για να επιληθούν. Αν σκεφτούμε λοιπόν τι μήνυμα θα θέλαμε να δώσουμε, έχουμε το παράδειγμα του Natura 2000. Αν το δούμε απ' έξω από την Ευρώπη, αυτό είναι ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό πλαίσιο πολιτικής καλύπτει 80% του, του εδάφους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύπτει ένα τεράστιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Σε αριθμητικό επίπεδο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν μας δίνει τα απαραίτητα αποτελέσματα. Φυσικά ο φορέας μας αντιμετωπίζει τη συμμόρφωση. Όταν υπάρχουν λοιπόν οι αναφορές που δίνουν τα κράτη-μέλη βάσει του άρθρου 17 και άλλων άρθρων. Παρακολουθούμε αυτά τα οποία κάνουν. Από όλα αυτά όμως προέκυψε και μια προειδοποίηση ότι ενώ είχε εφαρμοστεί η Natura 2000 η οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη μας, αυτό το οποίο δεν γινόταν ήταν να προστατεύονται τα άγρια είδη και τα ενδιαιτήματά τους. Όταν δούμε λοιπόν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων και την αξιολόγηση για την προστασία τους, βλέπουμε ότι σχεδόν το 1 τέταρτο των ζώων, είτε είναι αμφίβια, είτε είναι θηλαστικά, είτε είναι πλήνα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης. 62% των ε, διατημάτων και 50% όλων αυτών των πτηνών φαίνεται ότι βρίσκονται σε μία ε, αρνητική κατάσταση και πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ε, εξάλληψης και πάρα πολλά γνωστά εδιπτυνών έχουν μειωθεί οι αριθμοί τους. Επομένως, η διάγνωση αυτή που έχουμε μας λέει ότι ακόμα και αν κάνουμε τα σωστά πράγματα και έχουμε τις σωστές ε, περιοχές που γράφουμε στο χάρτη, αυτά τα οποία γίνονται δεν επιτυγχάνουν πράγματι τους στόχους μας. Τώρα, μα είναι δύσκολα τα προβλήματα και τα επιχειρήματα είναι περίπλοκα ένα από αυτά τα επιχειρήματα είναι το οικονομικό επιχείρημα. Ξέρουμε από τη μελέτη της Natura 2000 ότι τα ωφέλη που φέρνει αυτή η οδηγία στην Ευρώπη είναι της τάξης των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχει λοιπόν ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να κινητοποιήσουμε. Σε τοπικό επίπεδο αυτό που βλέπουμε είναι ότι είναι διαφορετικά τα δημοσιονομικά ε, μέσα που έχουμε, οι τρόποι με τους οποίους εμείς μπορούμε να εξηγήσουμε τι θα σήμαινε η απώλεια αυτών των περιοχών και των οικοτόπων και των ε, ζώων που ζουν εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια στην ε, τράπεζα αυτή δεδομένων μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία για τη χώρα σας, τι έχει κάνει, πώς έχει εφαρμόσει όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό το οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μια καλύτερη ε, η ιδέα του πώς θα αντεπεξέλθουν όλα αυτά τα στοιχεία, οι οικότοποι και τα άγρια ζώα και πτηνά με τις μελλοντικέ εξελίξεις. Και δεν λέω εδώ πέρα για πρόσθετες πιέσεις από τη γεωργία, αλλά ακόμα και με τα σημερινά σενάρια πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την απώλεια όλων αυτών των οικοτόπων και των αγρίων ειδών. Οι αλλαγές στο, στην ποιότητα των υδάτων, των της ατμόσφαιρας, η αλλαγή του κλίματος, όλα αυτά τα οποία συζητάτε στην Επιτροπή σα, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στα ίδια αυτά και τα οικοσυστήματα. Το φυσικό μας κεφάλαιο λοιπόν αυτή τη στιγμή <clears throat> χάνεται λόγω βιολογικών και φυσικών διαδικασιών και οι πολιτικές μας συγχρόνως δυσκολεύονται πάρα πολύ να παρακολουθήσουν αυτή την αλλαγή. Δεν προχωρούν αρκετά γρήγορα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και να επιτύχουν τους τελικούς στόχους. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Εμείς, εσείς ως νομοθέτες, έχετε την, το καθήκον της προστασίας και της εφαρμογής της νομοθεσίας, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να δείξουμε και μεγαλύτερη ευφυΐα. Γιατί η κατάσταση αυτή την οποία περιγράφω αφορά και την διάβρωση πραγματικής, πραγματικών στοιχείων αξίας για την οικονομία. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας πενθυμίσω την ε, σύμβαση του Όρχους και να σταθώ στο ρόλο των πολιτών. Σε πολλές χώρες η προστασία του περιβάλλοντος είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες. Έχουν ένα πάθος για τη φύση ή τουλάχιστον κατανοούν ότι το φυσικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να δούμε από τα αποτελέσματα. Δεν είναι τόσο εύκολο για την ποιότητα του αέρος, αλλά η φυσική οικότοπη είναι κάτι το οποίο είναι ορατό. Και μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κινητοποίηση των πολιτών. Αυτό γίνεται πολλές φορές σε εθνικό και υποεθνικό επίπεδο. Δεν έχουμε πάντα αρκετούς ανθρώπους για να αγωνιστούν. <clears throat> Νομίζω ότι η κινητοποίηση των πολιτών είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους με τους οποίους εσείς ως νομοθέτες μπορείτε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη επαγρύπνηση για το πώς γίνονται οι αλλαγές εμείς λοιπόν στο φορέα περιβάλλοντος έχουμε υποστηρίξει σε πολλές χώρες, τη Δανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ισπανία, τις απαρχές ενός παρατηρητηρίου πολιτών σε σχέση με την προστασία και την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και κυρίως για την προστασία από διαισθητικά ε, ξένα είδη. Αυτό το οποίο μας κοστίζει της τάξεως του των 20 δισεκατομμύριων ε, ευρώ το χρόνο. Είναι διάφορα φυτά και είδη τα οποία έρχονται από άλλες ε, υπήρους, αλλά σιγά σιγά μπαίνουν στο φυσικό περιβάλλον ανάμεσα στα ηθαγενή είδη. Επομένως η νομοθεσία για τα ε, επιθετικά, για τα φυτά, για, τα είδη τα οποία εισβάλλουν στο δικό μας περιβάλλον, εάν δεν εφαρμοστεί ουσιαστικά θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση πολλών άλλων μέτρων που λαμβάνουμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το οποίο θέλω να πω εν κατακλείδη είναι ότι η έλλειψη πληροφορίας δεν είναι δικαιολογία για την αδράνεια. Το κόστος της αδράνειας εδώ είναι ακόμα πιο μεγάλο από το κόστος της κλιματικής αλλαγής χωρίς το φυσικό περιβάλλον, χωρίς τα οικοσυστήματα, χωρίς την δυνατότητα να καθαρίσουμε τα ύδατα και την ατμόσφαιρα. Πολλά από αυτά που κάνουμε σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, με την αλλαγή της ενεργειακής σύνθεσης, ποιότητα υδάτων και ατμόσφαιρας δεν θα είναι, όλα αυτά δεν θα είναι εφικτά. Νομίζω ότι είναι η σύνδεση μεταξύ αυτών που φαίνονται κάπως ε, ε ακατανόητα όπως είναι η βιοπικιλότητα, η ύπαρξη του φυσικού μας περιβάλλοντος και όλων αυτών των πραγμάτων που μας δίνει δωρεάν η βιοπικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον, αυτό δεν γίνεται κατανοητό. να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας σημαίνει ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα στεγανά, να μην υπάρχουν αυτοί οι οποίοι προστατεύουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας, αλλά χωριστά από αυτούς οι οποίοι προστατεύουν τα εδάφη ή τα ύδατα ή την ενέργεια. Και πρέπει να κινητοποιήσουμε όχι μόνο του πολίτες, αλλά και τους ιδιοκτήτες γης, δασών, ε, γεωργούς και τα λοιπά και να προωθήσουμε την ιδέα μιας βιοπικιλότητας σε όλη την Ευρώπη, να μην έχουμε μια μονοκόμματη μονάχα αντιμετώπιση και νομίζω ότι η νομοθεσία που υπάρχει στο σχέδιο δράσης για τη βιοπικιλότητα δείχνει ότι αυτή η περιφερειακή διάσταση είναι μια που διάσταση που πρέπει να την υποστηρίξουμε και όχι να προσπαθούμε να έχουμε νομοθεσία ενό είδου για όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ήσασταν ε, πολύ ε, σε αυτά που μας είπατε. Ακούσαμε στατιστικές, τις ξέρουμε και από την ιστοσελίδα σας. Έτσι μπορούμε να μάθουμε περισσότερα και μάλιστα εδώ στην αίθουσα υπάρχουν και κάποιες από τις εκθέσεις σας. όσον αφορά την διαχείριση αποβλήτων κλπ. κλπ. Κάνω και εγώ διαφήμιση, γιατί εσάς σας άκουσα πολύ συγκρατημένη. Την κάνω εγώ του διαφήμιση. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, σχόλια. Το λόγο έχει αίθουσα. Α, πιο ντροπαλού σας βλέπω σε αυτό το κομμάτι της σημερινής μας συνεδρίασης από ότι στο προηγούμενο. So Πρώτος από την Ελλάδα, από την Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ελληνικής Βουλής. Η κυρία Θεοδόρα Αυγερινοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η εισήγηση την οποία ακούσαμε. Θα ήθελα καταρχάς να επαναλάβω το σχόλιο το οποίο έκανα στην πρώτη παρέμβασή μου σε σχέση με την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών αλλά και των επενδυτών για τις δυνατότητες οποίες έχουν για την αξιοποίηση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, Ραμσάρελα και των άλλων προστατευόμενων περιοχών ιδιαίτερης φυσικής σημασίας και φυσικής ομορφιάς είναι, υπάρχει μεγάλη σύγκρουση στα θέματα χρήσεων γης, στα θέματα γεωργίας, ε, αξιοποίησης ε, των περιοχών ως χώρων ανανεώσιμων ε, τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τουρισμού και πάει λέγοντας θεωρούμε ότι μπορεί να επέλθει μια κοινή χρήση όλων αυτών των χώρων και πλήρη αξιοποίηση των περιοχών Natura. Είναι κρίσιμο για την Ελλάδα, που έχει πάνω από 27% ε, του χώρου τη σε περιοχέ Natura, αλλά και για όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ειδικότερο θέμα όσον αφορά την προστασία των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίε έχουν πληγεί μετά από φυσικέ καταστροφέ. Μέχρι τώρα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πρόσθετα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, είναι κυρίω ανθρωπιστικού χαρακτήρα και όχι φυσικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση δηλαδή και τη υποβάθμιση τη φύση. Αναφέρομαι στο Ταμείο Αλληλεγγύη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένω θα έπρεπε να δούμε μέσα και στη νέα προγραμματική περίοδο μία ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία απευθύνονται για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών έτσι ώστε να επεκτείνονται ακόμα περισσότερο από ό,τι σήμερα και στην ανασυγκρότηση των φυσικών περιοχών. Θα σας ε, φέρω ως παράδειγμα ότι στην ε, Ελλάδα μετά από τις ε, φυσικές καταστροφές του 2007, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτίμησε την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος σε πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, η χώρα πήρε μόλις 2 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμα και σήμερα, 5,5 χρόνια μετά, δεν έχουμε αποκαταστήσει τις τα φυσικά μέρη και κυρίως τη Natura 2000 που έχουν υποβαθμιστεί από τις πυρκαγιές. Ε, δευτερευόντως, ήθελα να δώσω ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της θαλάσσιας βιοπικιλότητας, όπως ακριβώς αναφέρατε και εσείς. Το θέμα των ξένων, των ξενικών ειδών απειλεί τις περιοχές της θαλάσσιας βιοπικιλότητας και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο που είναι μια κλειστή θάλασσα. Το ίδιο και η υπεραλίευση αλλά και η παράνομη αλία. Το ίδιο και οι πηγές ρήπανσης τόσο από, την, από τα πλοία όσο και από τις πηγές από την ξηρά, κυρίως βέβαια η γεωργία. Θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση Τη ρήπανση και τη υποβάθμιση τη θαλάσσια βιοπικιλότητας, φαίνεται ότι αυτή τη, στιγμή, αυτή τη στιγμή και η Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουμε αξιοποιήσει τους πόρου που μας δίνει η θαλάσσια βιοπικιλότητα και είμαστε μπροστά στον κίνδυνο να την χάσουμε πολύ πριν μάθουμε όλα τα θετικά, είτε αφορά στα θέματα τη ιατρική, είτε στα θέματα τη ισορροπία του οικοσυστήματος, είτε γενικότερα τη υγεία και τη ζωή του ανθρώπου που μπορεί να μα προσφέρει η αξιοποίηση τη θαλάσσια βιοπικιλότητα. Πάνω σε αυτού του δύο άξονε, καταρχά, θα ήθελα να κάνω δύο προτάσει. Πρώτον, σε, στο θέμα τη διατήρηση βιοπικιλότητα εν γέννη, ε, εν ώψη και των φυσικών καταστροφών, να ενταθούν οι, προ, οι προσπάθειε, τα projects τα οποία έχουν να κάνουν με την αποτίμηση και τη διατήρηση τη βιοπικιλότητα, είτε στατικά μέσα σε τράπεζε βιοπικιλότητα, είτε σε πιο δυναμικά projects, και εμπλουτισμού της βιοπικιλότητας που τίνει να καταστραφεί λόγω ε, των φυσικών καταστροφών που έχουν επέλθει και βέβαια αυτό να λειτουργήσει προληπτικά και ε, εν ώψη και των κλιματικών αλλαγών τα οποία εντείνουν ακόμη περισσότερο του κινδύνου και την πίεση της που ασκούνται στη βιοπικιλότητα. Όσο δεν αφορά στην θαλάσσια βιοπικιλότητα, ίσως θα ήταν καλό από τώρα να σκεφτόμαστε κάποιου μηχανισμούς όπως ένα παρατηρητήριο για την διατήρηση της θαλάσσιας βιοπικιλότητας και για την ανάδειξή της, καθώς επίσης και τις ε, περιοχές προστασίας θαλάσσιας βιοπικιλότητας, όχι μόνο τι Ποσειδονίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά και τις περιοχές απαγόρευσης αλίευσης. Πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα τον, κλείνοντας να τονίσω και την ανάγκη ενδεχομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί τελικά και την υιοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ως ευρωπαϊκής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης για να προστατεύσει το θαλάσσιο περιβάλλον που βρίσκεται ή εν δυνάμει μπορεί να βρεθεί εντός αυτής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Σε το συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ στο πρώτο τμήμα αυτού του δεύτερου τμήματος, τι να κάνουμε, δημοσιογράφοι στην πολιτική ζωή μερικές φορές παίρνουν το πάνω χέρι. Α, ξεχάσετε το τηλέφωνό σας εδώ, κύριε Σουλτέ. Ε? Επόμενος ομιλητής είναι από τη Σουηδία. Ο κύριος Γέλμερετ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Βλέπουμε ποιε είναι οι φιλοδοξίε των χωρών μελών. Θέλω όμω εδώ να αναφέρω ότι εμεί στο Συνδικό Κοινοβούλιο έχουμε μία επιτροπή η οποία εξετάζει τους εθνικούς μας στόχους σε διάφορους τομείς. Έχουμε τους εθνικούς στόχους, έχουμε όμως και, τους, και τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αποφάσεις, όπως για παράδειγμα για το Natura 2000. Υπάρχουν και διεθνείς συμφωνίες από την άλλη μεριά. Κανονικά όλα αυτά θα έπρεπε να είναι αλληλένδετα. Μερικές φορές οι στόχοι όμως είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Είναι σε διαφορετικά επίπεδα περιβαλλοντικής προστασίας. Υπάρχει το κλίμα, υπάρχει η βιοπικιλότητα. Και από την άλλη θα έπρεπε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενσωματώσουμε τους στόχους έτσι ώστε να είναι πράγματι αποτελεσματικοί. Συγκρίνοντας με άλλες χώρες βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες που αντιδρούν τελείως διαφορετικά όταν μιλάμε για προστασία της φύσης. Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Υπάρχουν έξι, η Σουηδία και η Φιλανδία προστατεύουν 10% σε εθνικό επίπεδο, η Γερμανία 60% οι κατοχώρες 25%. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης. Η Σουηδία είναι πολύ περιοριστική όσον αφορά την προστασία των δασών, για παράδειγμα. Φυσικά και πρέπει να μάθουμε ημένα από τους δε όσον αφορά την επίτευξη στόχων. Να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα σωστό επίπεδο όμως, ώστε να μην υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στους εθνικούς και τους διεθνείς στόχους. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Έχω άλλους δύο ομιλητέ, την κυρία Εστρέλα και τον κύριο Φράγκο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν έχει ζητήσει κανείς άλλο το λόγο από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τέσσερι από τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν πήραν όμω το λόγο στον πρώτο γύρο νωρίτερα. Η κυρία Μπουρζάη, ο κύριος Γκορζίκα, η κυρία Σνόη και ο κύριος Άρκιτ. Αν κάποιο από αυτού του τέσσερι εξακολουθεί να θέλει το λόγο τώρα στο δεύτερο γύρο, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα όμω, η κυρία Στρέλα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου για αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα. Η ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα, κατά τη δική μου άποψη, έχει απασχοληθεί υπερβολικά με τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα και η συζήτηση αυτή που κάνουμε σήμερα μπορεί να συμβάλλει στο να επαναξισορροπηθεί με την εισαγωγή αυτού του τόσο σημαντικού θέματος για την προστασία του περιβάλλοντος. Όπως είπε και η κυρία Μακλέιτ, η προστασία της βιοπικιλότητας είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως μέσα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων στην κοινή αγροτική πολιτική και της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο προοπτικών θα πρέπει επίσης να δώσει να διαθέσει τους απαραίτητους πόρους <clears throat> για τη στρατηγική προστασίας βιοποικιλότητας με ορίζοντα το 2020 και αυτή η χρηματοδότηση θα αποσβεστεί ουσιαστικά από το ίδιο το περιβάλλον δεδομένου ότι μέχρι το 2050 η απώλεια βιοποικιλότητας και το κόστος της μπορεί να φτάσει στο 100% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη στιγμή το κόστος του Natura 2000 είναι 12 με 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Οι πολίτες μας λοιπόν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση για την Natura 2000, η οποία όμως συγχρόνως η χρηματοδότηση έχει σαν στόχο και να εξασφαλίσει την εφαρμογή των οδηγιών για τους οικοτόπους, για τα ε, ύδατα, για την θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και οι πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε σχέση με τις πράσινες υποδομές και η νομοθεσία που αφορά τα επιθετικά ξένα είδη τα οποία βρίσκονται στον, στο περιβάλλον το ευρωπαϊκό όπου οι προτάσεις Κομισιόν είναι πράγματι θετικές. Για να μπορέσω να κλείσω λοιπόν στο σημείο αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβαστούμε τους στόχους της ε, βιοποικιλότητος με φιλόδοξα σχέδια. Πρέπει όμως να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της κοινή γνώμη. Οι πολίτες μας θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η βιοποικιλότητα <clears throat> περιλαμβάνει όλες τις ε, αλληλεπιδράσεις μέσα στο γήινο οικοσύστημα και έχει να κάνει και με την ανθρώπινη δραστηριότητα, με την διατροφή, με την υγεία, με την ένδυση, με την ε, θέρμανση των κτίριων. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν επιπτώσεις στην ε, βιοπικιλότητα. Η βιοπικιλότητα είναι τελικά μια εγγύηση για την ανθρώπινη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος ε, θα ήθελε να πάρει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από τα Εθνικά Κοινοβούλια, του οποίου δεν έχω αναφέρει το όνομα. Έχετε το λόγο. Ε, dziękuję bardzo, panie przewodniczący Tadeusz Arkit. Θα Σας ευχαριστώ. Λέγομαι Τατέος Άκετ και εκπροσωπώ το Κοινοβούλιο της Πολωνίας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, στο Κοινοβούλιο της χώρας μου. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που συζητήσαμε. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα γιατί ό,τι κάνουμε όσον αφορά τη διαχείριση των υποβλήτων έχει άμεσες επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Πολωνία έχει πάρει πολύ σοβαρά την διαχείριση των ε, αστικών αποβλήτων και υπάρχει μία υπηρεσία η οποία παρακολουθεί ακριβώς αυτό το θέμα. Έχουμε εξάλλου υιοθετήσει μία νέα νομοθεσία και υπάρχει ένας χάρτης ε, βάσει του οποίου γίνεται η επεξεργασία και η διαχείριση των αποβλήτων. Και αυτό όχι μόνο γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την κοινοτική νομοθεσία, τους κοινοτικούς κανόνες, αλλά γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την προστασία του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά την ανακύκλωση κάποιων ε, ουσιών και κάποιων ε, υλικών που βρίσκονται στα απόβλητα, προσπαθούμε να επεξεργαστούμε με τον καλύτερο τρόπο αυτήν την πρώτη ύλη. Όπως μας είπε ο Επίτροπος, θεωρούμε και εμείς ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα οικονομική δραστηριότητα την οποία προωθούμε με δημιουργία δυνάμει πολλών θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό και επενδύουμε πολύ σημαντικά ποσά σε έργα υποδομών. Εν μέσω αυτής της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας της ε, κρίσης θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό επαναλαμβάνω και γιατί δημιουργούμε νέες θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και σας κυρία μου για την καλή σας παρουσίαση. Είμαι εισηγητής του 7ου προγράμματος πλαισίου για το περιβάλλον. Από αυτά που γνωρίζουμε, πιστεύουμε ότι είναι καλό να έχουμε ευρωπαϊκές διατάξεις, αλλά και να συνεργαζόμαστε σε διεθνή φόρο, όπως είναι το IPPS, για την βιοπικιλότητα. Πιστεύω επίσης ότι η συνεργασία με τις χώρες που γυτνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης ζωτική σημασίας. Για να έχουμε στοιχεία, για παράδειγμα για τα δάση, πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τις χώρες που βρίσκονται νοτίως της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Franco. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φράνκο. Άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Αν όχι, τότε Έχω μια τελευταία ερώτηση για σας κυρία Μαγκλέιτ, εγώ. Ήμουνα εισηγητής όσον αφορά τη στρατηγική και την βιοπικιλότητα. Και υπήρξαν κάποια πράγματα που με ξέπληξαν. Το ένα ήταν η σημασία που δίνουμε στο να ενσωματώσουμε την βιοπικιλότητα σε άλλους τομείς. Κοινή γεωργική πολιτική, για παράδειγμα, που καλύπτει το 50% του εδάφους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντική η γεωργία για την προστασία της βιοπικιλότητας. Τώρα που συζητάμε, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και χώρες μέλη, μειώνουν τελικά το πρασίνισμα της κοινή γεωργικής πολιτικής. Οπότε, ρωτάω, για σας ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά την προστασία της βιοπικιλότητας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι διαπιστώνω ότι ακόμη και στη δικιά μου τη χώρα, την Ολλανδία, όταν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν επικεντρωνόταν τόσο πολύ στην προστασία της φύση για να το πω έτσι ίδια, η ευρωπαϊκή δομή, αν μη τι άλλο, προσέφερε μεγάλη νομική βεβαιότητα για τους πολίτες. Γιατί υπήρχαν οι απαιτήσει όσον αφορά την προστασία της φύσης που μας ερχόντουσαν από την Ευρώπη. Αυτά. Παρακαλώ κυρία Μαγκλέιτ για να απαντήσετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από αυτή την τελευταία ερώτηση, η οποία βέβαια έχει επιπτώσεις και για τις άλλες. Όντω λέτε ότι οι πολίτε στρέφονται προ την Ευρώπη προκειμένου η Ευρώπη να προστατεύσει το τοπικό του περιβάλλον, την δικιά του φύση. Είναι μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει που αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί όλο και περισσότερο οι διαστάσει των προβλημάτων που από το τοπικό πάνε στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν σαν αποτέλεσμα να φεύγουν πέρα από την συζήτηση σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς γίνεται ο διάλογος. Μια από τις δουλειές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος πράγματι είναι να επιμένει στο σημείο αναφοράς. Είτε πρόκειται για το κτηματολόγιο. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει το πρόβλημα αν δεν έχετε καλά ορισμένα τα ε, δικαιώματα ιδιοκτησίας και αν ε, δεν είναι όλα αυτά αποσαφηνισμένα βάσει ενός κτηματολογίου, ποτέ δεν θα έχετε ένα ικανοποιητικό σύστημα προστασίας από τις πυρκαγιές. Μια λοιπόν από τις δικές μας δουλειές είναι να διασφαλίσουμε ότι τα όρια, τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία, το κτηματολόγιο, όλα αυτά να στέκουν μαζί. Γιατί αυτά είναι που θέλουν οι πολίτες, αυτά περιμένουν οι πολίτες, να δούνε πώς σε αυτά η Ευρώπη αντικατοπτρίζεται. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η κοινή γεωργική πολιτική και πώς αυτή φτάνει στο δικό μας στον αγρό, για να το πω έτσι απλά. Έχουμε δει ότι είναι πολύ δύσκολο η επιστημονική κοινότητα να μεταφέρει την γνώση που απαιτείται έτσι ώστε να πάμε από το παγκόσμιο ή το ευρωπαϊκό να κατέβουμε στο πολύ τοπικό. Τώρα είμαστε σε διαφορετική κατάσταση βέβαια από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Είναι δύσκολο πάντα όμως να δούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να την ερμηνεύσουμε πολύ συγκεκριμένα στο δικό μας το χώρο. Αν όμως υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι εθνικοί νομοθέτες πρέπει να την ενσωματώσουν με έξυπνο τρόπο στην πραγματικότητα που έχουν επιτόπου. αν δούμε όλες τις συζητήσεις που γίνονται για τον ορισμό προστατευμένων περιοχών. Από τη Σουηδία οι συνάδελφοί τι λένε, λένε ότι υπάρχουν τόσο πολλές ε, ε, περιοχές προστατευμένες, 685 τέτοιες περιοχές. Τι κάνουμε εμείς, προσπαθούμε να τις βάλουμε σε κατηγορίες, σε τρεις κατηγορίες. Μία που έχει να κάνει με την ε, διατήρηση, το δεύτερο που έχει να κάνει με τους τομείς, δηλαδή δάση, η παράκτια, τα δάση σε σχέση με τις πυρκαγιές, τα παράκτια σε σχέση με την αστικοποίηση. Είναι δηλαδή αυτή μια δουλειά που κάνουμε προκειμένου οι πολίτες μιας χώρας να μπορούν εύκολα να δούνε κατά πόσο η μεταχείριση που τους επιφυλάσσεται είναι δίκαια ή όχι, να μπορούν να συγκρίνουν επίσης. Και έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε σε διεθνείς συγκρίσεις να στηρίξουμε το IBBS ή ό,τι άλλη διεθνή συμφωνία υπάρχει. Αν εμείς δεν πάρουμε την δουλειά μας στα σοβαρά και δεν φροντίσουμε για αυτήν την ερμηνεία μιας νομοθεσίας από το ευρωπαϊκό, το κεντρικό επίπεδο στο τοπικό, ε, δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Τώρα αυτό το οποίο κάνουμε καλά είναι ότι έχουμε μια πολύ πλήρη ε, θα έλεγα δικτύωση και επιρροή στα δρόμενα σε διεθνές επίπεδο, είτε πρόκειται για την βιοπικιλότητα είτε άλλα. Δηλαδή πραγματικά μας αντιμετωπίζουν σαν τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, γιατί σε αυτά τα πράγματα έχουμε εναρμόνιση και ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Επ' αυτού λοιπόν η πρόοδος είναι μεγάλη. Όμως πώς οι συμφωνίες αυτές οι διεθνείς φτάνουν στο τοπικό επίπεδο, αυτό είναι λιγότερο σαφές. Τώρα γιατί, για αυτά που είπατε από την Ελλάδα, η διοπικιλότητα όντω είναι ο φτωχό ε, συγγενής. Είναι ένα θέμα πολύ ορφανό. Δεν έχουμε εξοδέψει αρκετό χρόνο και δεν έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες, πράγματι. Οι πολίτες όμως έχουν ένα ρόλο να παίξουν εδώ, είτε πρόκειται για τους αλλοίς, είτε πρόκειται για άλλους χρήστες της θάλασσας. Και έρχομαι τώρα και στα υπερπόντια διαμερίσματα που πολλές φορές τα ξεχνάμε. Πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ευθύνη για τις υπερπόδιες τους κτήσεις, όπου εκεί έχουμε τεράστια βιοπικιλότητα. Άρα πρέπει να προσέξουμε και να δώσουμε σημασία και σε αυτά που συμβαίνουν στα υπερπόντια διαμερίσματα, όπως και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου αυτής δεν μπορούμε όμως τώρα να αλλάξουμε το καθεστώς χρηματοδότησης ή τις πολιτικές. Αν δεν έχουμε κατανοήσει καλά, σε τοπικό επίπεδο, πώς έχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Είτε πρόκειται για τα απόβλητα, είτε πρόκειται για τη χρήση γης, είτε πρόκειται για τη δασοκομεία. Οι επιλογές που κάνουμε πρέπει να είναι ζωντανές. Και πάντα δίνω ένα παράδειγμα. Δανία. Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι επειδή εμεί βρισκόμαστε στη Δανία, αλλά είναι επειδή εκεί γίνονται πολλά. Η, η υπηρεσία μας, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, συμμετέχει στην ε, ε τοπογράφηση, στο κτηματολόγιο για τα ύδατα, τη γη, την βιοπικιλότητα, την ποιότητα του αέρος, δίκτυα που ζει ο κόσμος κλπ. Και το ότι επηρεάζουν όλα αυτά τη λήψη αποφάσεων έχει οδηγήσει σε πολιτικές, για παράδειγμα την προσαρμογή για το κλίμα, όπου προσπαθούμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις και να υιοθετήσουμε σωστά προγράμματα τον έχουμε ε, δεδομένα στο οποίο να μπορούμε να αναφερόμαστε και που τα έχουμε εμείς, αυτό πιστεύω ότι είναι μια από τις πιο πολύτιμες βάσεις δεδομένων που μπορεί να έχει κανείς και που μπορείτε και εσείς να χρησιμοποιήσετε. Αυτό το λέω και για την Πολωνία. Εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς οι διάφορες αποφάσεις διάζονται μεταξύ τους. Πάντως το νέο καθεστώς αδειοδότησης, η υπηρεσία για την προστασία και η υπηρεσία για την αδειοδότηση φυσικά και πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους. Αυτές είναι επιλογές που πρέπει να τεθούν και να τις γνωρίζει και ο κόσμος για να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς γίνεται. Ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο επίση προσπαθεί να στηρίξει τη δουλειά που κάνουν ε, και άλλοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράδειγμα, για την προστασία υδάτων. Δεν μπορείτε όμω να περιμένετε ότι μονομερό μπορούμε να βοηθήσουμε. Εμεί την ενημέρωση την κάνουμε. Ο κόσμος όμως πρέπει όχι μόνο να ενημερώνεται, αλλά να τον προσελκύει και η ενημέρωση αυτή. Υπάρχει μια εφαρμογή, μπορείτε να έχετε και στα τηλέφωνά σας, με την οποία ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί για την ηχορύπανση στην πόλη που ζει, για την ποιότητα των υδάτων εκεί που ζει. Και έχουμε εκατομμύρια επισκέπτες. Είναι σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει και να ενημερώνεται και να ενημερώνει για το τι συμβαίνει στον χώρο του. Και πάνω σε αυτό πρέπει να βασιστούμε για τις μελλοντικέ αποφάσεις και τη μελλοντική νομοθεσία. Ο κόσμος να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και διάδραση μαζί του. Οι πολιτικοί ιδιαίτερα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα να χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα στην καθημερινή του ζωή. Και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να συνδυαστεί και με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μακλέιντ. Πριν προσπαθήσω να φτιάξω κάποια συμπεράσματα, ο συνάδελφος από το Κοινοβούλιο της Σλοβενίας, ο κύριο Κόλο, έχει ζητήσει το λόγο. Θα σε ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενώσεις και σύλλογοι στην Σλοβενία που ανησυχούν όσον αφορά το εάν θα παραμείνει δημόσιο αγαθό το νερό. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ επίκαιρο και ακούγοντας ε, τις διάφορες προτάσεις για τη νέα νομοθεσία, οι ανησυχίες αυτές ε, επανέρχονται. Θα ήθελα επίσης να πω ότι όσον αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ε, βιοπικιλότητα και αυτό σε επίπεδο εκπαίδευσης και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πολύ πολύτιμες αυτές οι παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω και εγώ να προσθέσω κάποια συμπεράσματα. Καταρχήν, ευχαριστώ όλους σας για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Έχουμε 13 προέδρους και αντιπροέδρους επιτροπών από τα Εθνικά Κοινοβούλια, μέλη των Επιτροπών Περιβάλλοντος, των Εθνικών Κοινοβουλίων, πολυάριθμους συναδέλφους δηλαδή από τα Εθνικά Κοινοβούλια και πολλές φορές όταν ε, ακούμε τέτοιου είδους συζητήσεις ακούμε τις προτάσεις υπέρ ή κατά της ε, Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Αυτό που διαπιστώνω όταν συζητούμε για το περιβάλλον και ασχολούμαι αυτά τα θέματα από το 1992, διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο. Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια υπάρχουν πολύ ισχυρές προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της φύσης η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών σε αυτή τη συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική στον τομέα του περιβάλλοντος και της φύσης. Εδώ έχουμε την Επιτροπή Αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επεξεργάζεται αναφορές από τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αυτών των αναφορών που έχουν σαν θέμα το περιβάλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι η συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών είναι πολύ μεγάλη για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό και ο δικός σας ρόλος είναι πολύ σημαντικός στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική λοιπόν η σημερινή μας συνάντηση και νομίζω ότι αναφερθήκαμε σε θέματα που αφορούν το νερό, τα απόβλητα, την προστασία του περιβάλλοντος σε διασυνεργικό επίπεδο, με πολύ υψηλό επίπεδο ομιλητές που έκαναν παρατηρήσεις χρήσιμες, επικοδομητικές. Ακούσαμε πολλές πλευρές, ακούσαμε την ανησυχία πολλών ομιλητών για το πώς μπορούμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη συμμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ιδιαίτερα με ικανοποίησε το γεγονός του ότι αναφερθήκατε πολλές φορές σήμερα το απόγευμα σε μέτρα που αφορούν φορολογικά κίνητρα. Επίσης στα διάφορα επίπεδα, το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό, το τοπικό, οι επιχειρήσεις, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι στο μέλλον η βιώσιμη ανάπτυξη σίγουρα θα στηριχθεί από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και όχι από τις κυβερνήσεις. Υπάρχει λοιπόν πολύ δυναμικό και πολλές δυνατότητες από μέρους των επιχειρήσεων. Καλύτερη λοιπόν συνεργασία, διασυνοριακή συνεργασία και βεβαίως η σημασία του να συνειδητοποιήσει η κοινή γνώμη. Σας ανέφερα ήδη το παράδειγμα της Επιτροπής Αναφορών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ενδιαφέρον των πολιτών που καθημερινά αυξάνεται. Κάποιοι αναφέρθηκαν επίσης στο θέμα της ολοκληρωμένης ε, πολιτικής τη συμμετοχή της, ε, του περιβάλλοντος σαν συνιστόσα όλων των άλλων πολιτικών, το θέμα της ε, αλλιευτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε περισσότερο στην γεωργία. Εδώ οι απόψεις ε, μπορεί να μην είναι κοινέ, αλλά έχουμε το θέμα της πράσινης γεωργίας, της πράσινης οικονομίας, κάτι που το υποστηρίζουν όλοι. Και κάτι που θα πρέπει να προχωρήσει όπως έγινε και στον τομέα της αλίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ για άλλη μια φορά, όπως το έκανε και ο Επίτροπος, στο κόστος που απορρέει από την μη συμμόρφωση, την μη εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και για τα απόβλητα οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, ένας ολόκληρος ε, βιομηχανικός τομέας που θα αποφέρει δισεκατομμύρια ευρώ και την δημιουργία πολλών χιλιάδων θέσεων απασχόλησης. Η Επιτροπή πιστεύει πραγματικά ότι εδώ μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και σε 400.000 νέες θέσεις απασχόλησης. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε με αυτά τα σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τέτοιες συναντήσεις, αλλά και με πιο σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας σε καθημερινό επίπεδο. Πρέπει να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, πρέπει να συνεχίσουμε την συνεργασία μεταξύ των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μιλάμε για έναν τομέα της πολιτικής που είναι ευρωπαϊκός, το περιβάλλον, σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε πολύ σύντομα και σας προσκαλώ όλους στο κοκτέιλ έξω από την αίθουσα όπου μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας πιο άτυπα και ανεπίσημα. Σας ευχαριστώ πολύ.